Hyvää Καλθίστε παρακαλώ, καλή σας μέρα και φορέστε τα ακουστικά σας για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε. Χθες το βράδυ είδαμε μία ταινία συμμετοχή των μητέρων του Τιάνναν Μεν. Και θα προχωρήσουμε σήμερα με την ακρόαση για θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Κίνα. Ο λόγος είναι ότι στις 24 ε, Νοεμβρίου διεξήχθη διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας και χθες έγινε και διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας και υπενθυμίζω ότι η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πάντοτε προσπαθεί να διασφαλίσει ώστε τα αποτελέσματα των διαφόρων διασκέψεων ή τα, διαφο τα αποτελέσματα μάλλον των συζητήσεων μας εδώ να φτάνουν εν τέλει μέχρι το επίπεδο των διασκέψεων. Για σήμερα έχουμε διαφόρους αγορητές. Έχουμε χρόνο μέχρι τις 11 για την συζήτηση αυτή. Πρώτα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μας δώσουν μια επισκόπηση του διαλόγου, των όσων διεξήχθησαν στο διάλογο και μετά θα ζητήσω από τους άλλους ομιλητές να λάβουν τον λόγο. Βέβαια θα, είναι και, ε, θα ακολουθήσει και συζήτηση που πιστεύω θα είναι ζωηρή. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τους συναδέλφους μας διότι ορισμένου από του θα, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από του προσκεκλημένου μα εννοεί η Πρόεδρο, διότι ορισμένοι από του συναδέλφου έρχονται με κάποια καθυστέρηση. Έχουμε τώρα εκπρόσωπο τη ε, Σουηδική Προεδρία, τον ε, πρέσβη κ. Νόρλαντερ, ο οποίο ε, θα μα εξηγήσει περί του ε, διαλόγου. Έχετε το λόγο κύριε πρέσβη. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εύχομαι καλημέρα σε όλου Θα ήθελα να αρχίσω με το νομικό σεμινάριο το οποίο προηγείται συνήθως του διαλόγου και όπως γνωρίζετε γίνεται πριν από τον διακυβερνητικό διάλογο. Τα θέματα ήταν αυτή τη φορά πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στην οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Είναι παρόν και ο καθηγητής Σέβας και θα μπορέσει να εξηγήσει περισσότερα για το σεμινάριο και την έκβασή του. Δεν θα ασχοληθώ λοιπόν εγώ περισσότερο με αυτό. Πάντως μας ικανοποίησε το ότι διεξήχθη το σεμινάριο. Είχαμε ορισμένα προβλήματα συμμετοχής. Εξάλλου κάνουμε και επίσκεψη επιτόπου όταν είμαστε στην Κίνα. Την φορά αυτή δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε με τους Κινέζους οικοδεσπότες σχετικά με τον τόπο που θα γινόταν η επιτόπου επίσκεψη. Έτσι, αντί να βγούμε εκτός Πεκίνου, επισκεφθήκαμε διάφορες κυβερνητικές αρχές και άλλες οργανώσεις, το ίδιο το Πεκίνο. Διεξαγάγαμε ενδιαφέρουσε συζητήσεις με πανεπιστημιακούς που ασχολούνται με την ομολογία, αλλά και με συνηγόρους υπερασπίσεως. Και συναντηθήκαμε και με εκπροσώπους κυβερνητικών ε, υπηρεσιών που ασχολούνται και με την τεχνική υποστήριξη και συνεργασία. Τα θέματά μας ήταν κράτος δικαίου, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, νομικές μεταρρυθμίσεις, ο ρόλος των συνηγόρων υπερασπίσεως και το θέμα της κράτησης χωρίς δίκη. Στην ημερήσια διάταξη αυτή και όχι μόνο στο σεμινάριο, υπήρχε και ένα θέμα για την ε, προώθηση και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων μέσα σε πλαίσια οικονομικής κρίσης, για το οποίο θέμα δεν υπήρξε επαρκής χρόνος. Και υπήρχε και το διαρκές θέμα της συνεργασίας σε διεθνείς οργανισμούς. για το ε, Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά και για τη συνεργασία με του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι Κινέζοι προσήλθαν με μεγάλη αντιπροσωπεία που εκπροσωπούσε πολλά υπουργεία και άλλους κυβερνητικούς οργανισμούς. Η ατμόσφαιρα στη διάρκεια των συνομιλιών ήταν καλή, όπως αναφέρουμε και στο ανακοινοθέν τύπου, ε, προχωρήσαμε σε ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θέσαμε το θέμα της κύρωσης από πλευράς Κινέζων την κύρωση δηλαδή της συνθήκης για δικαιώματα του πολίτη και ανθρώπινα δικαιώματα. Η διαδικασία αυτή της κύρωσης ε, υπάρχει εδώ και 10 χρόνια. Θέσαμε και το θέμα της θανατικής καταδίκης. Επ' δεν υπάρχουν νέα, παρότι ως γνωρίζετε υπάρχει μείωση του αριθμού των εκτελέσεων αφής το Κινέζικο Ανώτατο Δικαστήριο επανήλθε στην ε, επανεξέταση θανατικών καταδικών που έχουν αποφασίσει χαμηλότερου βαθμού δικαστήρια. Επανήλθαμε στο θέμα των μαύρων φυλακών. Πρόκειται για θεσμούς εντό εισαγωγικών χωρίς νομική βάση, όπου κρατούνται πρόσωπα χωρίς ε, δίκη και την ύπαρξη των οποίων αρνούνται οι Κινέζοι. Μιλήσαμε για θέματα ρόλου συνηγόρων υπερασπίσεως, για τις ταραχές που σημειώθηκαν στην Σινγιάνγκ και στο Θιβέτ. Όπως ξέρετε, η κινέζικη πλευρά θεωρεί ε, τις ε, ταραχές αυτές ως εγκληματικού χαρακτήρα και δεν ικανοποιήθηκαν με τα ανακοινοθέντα που είχαν εκδοθεί από πλευράς Ευρωπαϊκής πριν από τον διάλογο αυτό. Δηλώσεις δηλαδή οι οποίες κατεδίκαζαν τις θανατικές καταδίκες που επιβλήθηκαν σε πρόσωπα τα οποία είχαν ανοιχθεί στις ταραχές αυτές. Εν τέλει θέσαμε το θέμα του κράτους δικαίου, διότι διαπιστώσαμε ότι εμείς βλέπουμε μια επιδίνωση στην εφαρμογή κράτους δικαίου. Βλέπουμε ότι ένας αριθμός δικηγόρων στερήθηκαν την άδεια άσκηση επαγγέλματος, τους αφαιρέθηκε η άδεια άσκηση επαγγέλματος και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει και διορισμός ενός αριθμού αρχιδικαστών οι οποίοι στερούνται νομικής εμπειρίας. Και υπάρχουν και άλλα θέματα σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης. Από πλευράς της η Κίνα επέκρινε την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πλείονες χώρες μέλη της Ένωσης και στην Σουηδία, όπου τέθηκε το θέμα της κατάστασης των Σάμι και ε, σε σχέση με ένα τζαμί στην Νότια Σουηδία. Θα επανέλθουμε βεβαίως, θα δώσουμε γραπτές απαντήσεις ε, στους Κινέζους για τις κατηγορίες αυτές. Από την κινέζικη πλευρά λάβαμε γραπτές απαντήσεις για τις ατομικές περιπτώσεις τις οποίες είχαμε θέσει υπόψη τους και αυτό είναι καλό. Μετά το πέρας του διαλόγου κάναμε επίσκεψη αυροφροσύνης στον Υφυπουργό Εξωτερικών. Συζητήσαμε πάλι θέματα όπως η θανατική καταδίκη, όπως ε, η ε, συνεργασία με τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ο ίδιος ο Υπουργό δήλωσε ότι θεωρεί τον διάλογο σημαντικό μέρος των σχέσεών μας. Και για να προχωρήσουμε και ένα βήμα πιο ψηλά, η διάσκεψη έλαβε χώρα και στην διάσκεψη τέθηκαν πλήωνα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα οποία απηχούνται και στο ανακοινωθέν τύπου. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ετέθηκαν αλλά και, στο υπουργό των στο... και σε επίπεδο μάλλον συγγνώμη, Υπουργών των Εξωτερικών, αλλά με περισσότερες λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ ε, πολύ κύριε Πρέσβη. Ακούσαμε και πάλι ότι είναι πολύ σημαντικό να εξετάζει κανείς τον διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το πώς είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα εδώ στην Ευρώπη, γιατί και εδώ έχουμε ορισμένα προβλήματα. Και αυτά τίθενται στην διάρκεια του διαλόγου. Ένα σημαντικό θέμα, κύριε Πρέζη. Θέσατε το θέμα του Χουτζι Γιάνγκ που βραβεύτηκε πέρσι με το βραβείο Ζαχάροφ. Γνωρίζετε αν είναι ακόμη στην φυλακή και ποια είναι η κατάσταση της οικογένειάς του. Θέσαμε το θέμα αυτό, καθώς και άλλες ατομικές υποθέσεις που ξέφευγαν και από την λίστα την οποία είχαμε υποβάλει. Από την κινέζικη πλευρά δεν υπήρξαν απαντήσεις, εκτός από κάποιες τυπικότητες δηλαδή θέματα όπως πότε εκδόθηκε η απόφαση του δικαστηρίου και διάφορα τέτοια, αλλά δυστυχώς καμία λεπτομέρεια. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα τώρα να ακούσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Μιχάλης Ρόκας και ο Τόμπι Κίνγκ είναι παρόντες εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Λίγα έχω να συμπληρώσω στα όσα είπε ο κύριος Πρέσβης. για τον Χούτζια. Έχουμε κάποιες οφορίες, αλλά όχι από την κινέζικη πλευρά. Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση της υγείας του παραμένει επισφαλής, παρόλο που λαμβάνει τα φάρμακά του, αλλά παρόλα αυτά η υγεία του είναι έφραστη και αυτό μας ανησυχεί. Σε ό,τι αφορά την γυναίκα του, μάθαμε από διάφορες πηγές ότι είναι, έχει μεγαλύτερη ελευθερία τώρα είναι λιγότερο περιορισμένες οι κινήσεις της, παρότι όταν επισκέφθηκε την Κίνα ο πρόεδρος Ομπάμα, η γυναίκα αυτή τέθηκε υπό περιορισμό κατοίκων. Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο θέτουμε σε κάθε ευκαιρία. Τώρα, για την ίδια τη διάσκεψη κορυφή εκδόθηκε κοινό ανακοινοθέν. Χθε εκδόθηκε, υπάρχει μια παράγραφος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η υπαριθμόν 8, που είναι καλά διατυπωμένη μιλούμε για την κοινή δέσμευση για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, το κράτος ε, δικαίου, την ε, ε, πρόθεση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επίσης, επιβεβαιώνουμε και πάλι την υψηλή αξία που αποδίδουμε στον διάλογο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το σχετικό σεμινάριο και μια σαφής δέσμευση να συνεχίσουμε να, εργαζόμαστε, να συνεργαζόμαστε για να επιτελεστεί διαρκής πρόοδος. Τώρα για θέματα κύρωσης της ICCPR στην διάσκεψη επανεπιβεβαιώθηκε η δέσμευση να κυρωθεί. Αλλά βέβαια υπάρχει ανησυχία λόγω της καθυστέρησης των 11 ετών και αυτό δηλώθηκε καθαρά. Επίσης η ανάληψη υποχρέωσης συνεργασίας με τους μηχανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην διάσκεψη ε, κορυφής τέθηκαν. Τέθηκαν επίσης και από την Τρόικα, όπως είπε και ο κύριος Πρέσβης προηγουμένω, αλλά τα έθεσε και ο ίδιος ο πρόεδρος Μπαρόσο όταν ε, συναντήθηκε με Κινέζους ηγέτες, έδωσε και ιδιαίτερη έμφαση ε, στην συνεχιζόμενη αξιολόγηση του διαλόγου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όταν θα είμαστε έτοιμοι να επανέλθουμε θα είμαστε σε θέση να παραγάγουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτές τις λίγες συμπληρώσεις μονάχα είχα για τα όσα είπε ο κύριος Πρέσβης. Σας ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. πρόεδρος. Βέβαια, γνωρίζουμε σαφώς ότι το Συμβούλιο γνωρίζει τα σχετικά με τον διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε την έκθεση και σύντομα μάλιστα, ώστε να μπορέσουμε να γνωρίζουμε ποια είναι τα μέρη εκείνα του ε, διαλόγου ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω. Ας συνεχίσουμε τώρα. Έχουμε μια ε, αξιόλογη σειρά προσκεκλημένων εδώ κοντά μας. καλωσορίζει τον κύριο Γκάου που εκπροσωπεί τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα. Είναι ε, Senior Policy Advisor και έχει έρθει από τη Νέα Υόρκη για να μιλήσει σήμερα μαζί μας. Μας έχει υποβάλει μια ε, πλήρη ε, παρουσίαση, γραπτός, και θα ήθελα να σας παρακαλέσω αγαπητέ κύριε να θέσετε υπόψη μας τα βασικά σημεία της γραπτής παρουσίασης, ώστε να μείνει επαρκής χρόνος για συζήτηση μετά. Κύριε Γουανκιάο, έχετε το λόγο. Thank Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Μέλη της ε, Υποεπιτροπής, ευχαριστώ και εσάς για την ευκαιρία που μου προσφέρετε να συμβάλλω σε αυτήν την ε, συζήτηση τόσο επίκαιρη. Το σημαντικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ε, Κίνα, δικαιώματα των μειονοτήτων και εφαρμογή της ε, θανατικής ποινής που εκδόθηκε στις 25 Νοεμβρίου, καταγράφει με ακρίβεια και δείχνει τον κατεπήγοντα χαρακτήρα των προβλημάτων των σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα σήμερα αποστέλει το, το ψήφισμα αυτό ένα πολύ σημαντικό μήνυμα στην κινέζικη κυβέρνηση, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη, αλλά και ένα μήνυμα αλληλεγγύης και ελπίδας προς τον κινέζικο λαό. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω αφηγούμενο στην προσωπική μου ιστορία. Ήμουν ε, ερευνητής εντεταγμένος με στο σύστημα του Κομμουνιστικού Κόμματος για περισσότερο από 14 χρόνια, όταν ε, πριν από 20 χρόνια ε, ήμουν ε, μάρτυρας της αιματηρής καταστολής των κινημάτων της 4ης Ιουνίου στην πλατεία στην πλατεία Τιανανμέν και τότε απεκόπηνα από το σύστημα εξοριστικά και επειδή, δημοσιεύτηκα, επειδή δημοσίευσα το βιβλίο Zoo Lies ε, και τα τελευταία, τα τελευταία χρόνια του Zoo Lies που απογορεύτηκε από, το κινέζικο, από την κινέζικη κυβέρνηση μου απαγορεύτηκε η επιστροφή στην ε, Κίνα και δεν μπόρεσα ούτε τη μητέρα μου να δω πριν ε, ξεψυχήσει. Πλην όμως δεν είμαι εγώ μόνος σε αυτά τα προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά τα, και τις δύσκολες προσωπικές επιλογές, Επιλογέ που έχουν να κάνουν με τη συνείδηση, με τις αρχές που έχει ο καθένα ορίσει για τον εαυτό του και το ακριβό τίμα που καλούμαστε να πληρώσουμε, το έχουμε πληρώσει πολύ και το πληρώνουμε κάθε μέρα στην Κίνα. Καθώς ε, προβλήθηκε η ταινία για τις ε, μητέρες της πλατείας Τιερερμέν βλέπουμε πολλά παραδείγματα ανθρώπων που αγωνίστηκαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και που αγωνίζονται ακόμη κατά της ε, αμνησίας ως προς την ιστορία, ως προς της, ε, την, αγωνίζονται κατά της αποδοχής ενός τελεσμένου. και που αγωνίζονται για περισσότερο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα και συγκεκριμένου μηχανισμού και διαδικασίε. Θα ήθελα τώρα να μιλήσω λίγο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα. Μπορεί το θέμα των Ολυμπιακών, τη Ολυμπιάδα του 2008, να είναι ακόμη νοπό στη μνήμη μα, ωστόσο είναι αναμφίβολο. Όσο και αν αυτό το θέαμα προσπάθησαν να το καταστήσουν επίδειξη δυνάμεων της Κίνας, είναι αμφίβολο ότι το καθεστώς της Κίνας σήμερα είναι ένα καθεστώς το οποίο απλώς ε, επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις εις βάρος οποιοδήποτε επικρίνει την κυβέρνηση ή που απλώς όταν ε, υποδεικνύει ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. ή ενδεχομένως ε, διατυπώνει παρατηρήσεις οι οποίες μπορεί να μαυρώσουν την εικόνα του Κομμουνιστικού Κόμματος in the lead of 18th National Congress of the CPC in 2012. Ύστερα από το 18ο συνέδριο του κόμματος, Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας το 2012, μάλλον εν ώψη του Μεγάλου Συνεδρίου το 2012, ε, γίνεται μια διαλκυστίνδα μεταξύ διαφόρων παρατάξεων της, ε, του κόμματος για το ποιος θα κερδίσει την ε, εξουσία, ποιος θα πάρει το πάνω χέρι. Και βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ένταση και σκληρή γραμμή ε, σε επίπεδο και κυβέρνηση που προσπαθεί να ελέγξει το λαό αντί να αντιμετωπίσει τα θεμελιώδη προβλήματα. Ταυτόχρονα σημειώνονται πολύ σημαντικά προβλήματα ανασφάλειας σε επίπεδο ηγεσίας, ενώ η ε, διεθνής κοινότητα κατά βάση επιτρέπει στην Κίνα να δρά ανεξέλεγκτη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα ανεξέλεγκτα. Μόνο και μόνο γιατί οι ορισμένε κυβερνήσει θέλουν να διαφυλάξουν τι επενδύσει και τα συμφέροντά του. Ιδιαίτερα την πρόσβαση στην Κίνα, τι συναλλαγέ, το εμπόριο και θέματα ασφάλεια. η επέκταση αυτή τη στιγμή της ε, ήπιας λεγόμενης δύναμης της Κίνας αντανακλάται στις ε, ε, εκδηλώσεις που γίνονται σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, εκδηλώσεις όπου τιμάται η, η παράδοση, ο πολιτισμός της Κίνας. Αντανακλάται επίσης στα Ινστιτούτα Κονφουκιανισμού που πολλαπλασιάζονται στις πολιτιστικές ανταλλαγές. Με, βάση λοιπόν ε, πανεπιστημιακές ε, ή πολιτιστικές ανταλλαγές, αυτές οι πρωτοβουλίες της λεγόμενης ήπιας δύναμης αποτελούν ταυτόχρονα μια στρατηγική που υποστηρίζουν ε, οι επίσημες αρχές για την προαγωγή ενός κινέζικου μοντέλου, την προαγωγή της συνένεσης του Πεκίνου μέσω των επίσημων μέσων ενημέρωσης. Η διεθνή κοινότητα λοιπόν αποδεχόμενη αυτές τις επιδείξεις ήπια δύναμη, ουσιαστικά πέφτει στην παγίδα της ε, ε, αυταρχικής διακυβέρνησης του Κινέζικου Κομμουνιστικού κόμματο, το οποίο προσπαθεί να πει στον κόσμο ότι η Κίνα είναι μια έννοια, μια παράδοση, έχει ένα πολιτισμό διαφορετικό, κατά βάση διαφορετικό από τη Δύση και ω εκ τούτου θα πρέπει να εξαιρεθεί από την υποχρέωση σεβασμού των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με το να χορηγείται λοιπόν εν επιταγή στην Κίνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή με το να ε, κοφεύουν ε, οι υπόλοιπε χώρες στις φωνές των ε, ταραχοποιών από την Κίνα, ε, εντός εισαγωγικών ταραχοποιών, η διεθνής κοινότητα ουσιαστικά συμβάλλει στο να υπονομευθούν οι αγώνες των Κινέζων, μέσα και έξω από την Κίνα. Πρόκειται για επιλογές ή αν θέλετε ανταλλάγματα που υποβαθμίζουν ταυτόχρονα, υπονομεύουν ταυτόχρονα το διεθνέ σύστημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά μπορεί να έχουν και πολύ επικίνδυνε ε, συνέπειε ω προ την ευημερία και την ασφάλεια σε ολόκληρο τον κόσμο. Όταν, κάθε, όταν μια κυβέρνηση κάνει την επιλογή ε, του να παραγνωρίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, έναντι ε, κάποιου κέρδους εμπορικού ή σε όρους ασφάλειας, ε, ταυτόχρονα υπονομεύει και τα συμφέροντα, τα εσωτερικά. Επιδεινώνεται δηλαδή η κατάσταση και στην Κίνα, αλλά και στην εν λόγω χώρα, όπως και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η πολιτική που ακολουθεί η Κίνα για ε, υποβαθμισμένα ανθρώπινα δικαιώματα όπως και υποβαθμισμένα ε, δικαιώματα των εργατών αποτελεί και μια μεγάλη πρόκληση για την παγκόσμια οικονομία. Και τώρα θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια, αν μου επιτρέπετε, για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί κανείς ε, να ισχυριστεί ότι αντιλαμβάνεται τις διαδικασίες των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, τη λειτουργία τους ε, και ε, τον τρόπο με τον οποίο στέκονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, εάν συγκρίνει τη συμπεριφορά αυτή ε, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου και σε σχέση με την Κίνα. Ο διάλογος λοιπόν, η ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και τα σεμινάρια είναι πολύ χρήσιμες μέθοδοι και θα θέλαμε να ακούσουμε και στην σημερινή ευκαιρία τις απόψεις των άλλων ειδικών. Ωστόσο, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη πρέπει εν τέλει να αποστείλουν ένα συνεπές μήνυμα, ένα στεναρό μήνυμα στις κοινωνικές αρχές σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του ατόμου, τα δικαιώματα του ανθρώπου. Τις αρχές ε, τις οποίες έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμπεριλάβει ε, ως προϋποθέσεις για κάθε συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας στις διεθνείς, σχέσεις, διεθνείς σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω ήδη ε, λάβει μέρος και σε άλλα σεμινάρια, πέντε το, τα τελευταία οχτώ χρόνια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βλέπω ότι κάθε προσπάθεια για την προαγωγή των ανθρώπινων δικαιωμάτων ε, μέσα σε κάθε νέο τομέα ανάπτυξη πολιτικής, το λεγόμενο benchmarking, benchmarking το οποίο σημαίνει ε, εξέταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και εν ώψη κάποιες ε, εμπορικής ε, σχέσης νέας που συνάπτεται με άλλο κράτος, αποτελεί μια πολύ χρήσιμη μέθοδο. Δυστυχώς όμως δεν καταγράφεται στην υπόθεση αυτή ε, πρόοδος συγκεκριμένα πρακτικά αποτελέσματα τα οποία θα μπορούσε κανείς να επιδείξει. Το μόνο που υπάρχει είναι η ανταλλαγή απόψεων, ο διάλογος ο λεγόμενος και κάποια σεμινάρια Όλα αυτά υπό τον τίτλο της πολιτικής ανταλλαγής απόψεων ε, χωρίς δηλαδή καμία πίεση. Το ότι δεν αμφισβητείτε, δεν ε, ελέγχετε η ε, λογοκρισία στην Κίνα, το ότι δεν ε, αντιδρά κανείς το γεγονός ότι κάποιος επιλέγει ποιος θα έρθει να μιλήσει και το τι ακριβώς θα πει, αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Είναι ένα ε, μέσο που χρησιμοποιεί το status quo στο Πεκίνο η κυβέρνηση και συνεχίζει με τον τρόπο αυτό να παραβιάζει τα δικαιώματα του ανθρώπου. τα οποία ε, υποτίθεται ότι θα έπρεπε να προστατεύει. Η κυβέρνηση, όπως θα προβλέπει ε, η νομοθεσία της Κίνας και όπως θα έπρεπε να προαγόνται και μέσα στο διεθνή διάλογο, γιατί αυτά είναι υποχρεώσεις της Κίνας. Και κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω κάποιες συστάσεις. Καταρχάς, τα διάφορα ε, θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να υποστηρίξουν πιο αποτελεσματικά τις προσπάθειες των ε, Κινέζων αγωνιστών ε, για τα δικαιώματα του ανθρώπου. καθώς και του Διεθνού Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Κίνας, ε, το HRIC, καθώς εμείς συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για, περισσότερο, για πιο ανοιχτή κοινωνία, για περισσότερο διάλογο. Θα θέλαμε λοιπόν την υποστήριξή σας και θα θέλαμε επιπλέον περισσότερη διεκδίκηση λογοδοσίας για το παρελθόν. Δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ερετό δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα μπορεί να ασκήσει την εποπτεία του και την παρακολούθηση που δικαιούται να έχει στον τομέα των ανθρωπινών δικαιωμάτων, έτσι ώστε αυτά να επαληθεύονται σε κάθε περίπτωση ανάπτυξη πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό όρους λογοδοσίας και διαφάνειας. Ως προς το που ε, διατίθενται οι περιορισμένοι ούτως ή άλλως πόροι και τα ε, κονδύλια που προκύπτουν από, την εισφορά του Ευρωπαίου Φορολογουμένου. Ως προς τα σεμινάρια των εμπειρογνωμόνων, εάν τα σεμινάρια χρηματοδοτούνται από ένα μέσο δημοκρατίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου, θα πρέπει αυτά να αξιολογούνται και ως προς τα αποτελέσματά τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τι προσφέρουν δηλαδή. Εάν είναι απλώ ανταλλαγή απόψεων μεταξύ πανεπιστημιακών, μεταξύ ειδικών επιστημόνων, ε, θα προτείναμε να τηρηθούν οι προδιαγραφές που ισχύουν σε όλο τον κόσμο για την επιστημονική έρευνα, την ανεξαρτησία και την ακαιρεότητα μιας μελέτης. Αγωνιζόμαστε το HRIC και το FIDH ε, για να καταστήσουμε δημόσια την, ε, την εκτίμηση την οποία διατυπώσαμε το Δεκέμβριο του 2008 για τον διάλογο ως προς τα δικαιώματα του ανθρώπου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας και την ανάπτυξη ενός σεμιναρίου νομικών εμπειρογνωμόνων. Αυτή η εκτίμηση προτείνει συγκεκριμένες συστάσεις για την ενίσχυση διαφάνειας και της λογοδοσίας του μέσου και την ενίσχυση του ρόλου και της συμμετοχής ανεξαρτών με κυβερνητικών οργανώσεων ειδικοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το, με ειδικούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προτείνουμε λοιπόν να καταστεί αυτό, αυτή η μελέτη ε, μέρος των πρακτικών της ακρόασής σας. Και κλείνοντας, εάν δεν σημαίνουν τίποτα οι λέξει δικαιώματα του ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε τα κάτι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη θα πρέπει, μάλλον εάν έχουν κάποιο νόημα οι όροι δικαιώματα του ανθρώπου, τότε θα πρέπει να αναλάβουν συγκεκριμένα μέτρα τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να τα σεβαστούν. Η Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βουέγγιαν Γκάου, ήταν πολύ εύστοχε οι παρατηρήσει σα. Πρόκειται για ζητήματα τα οποία διαρκώ υποβάλλουμε εμεί στο Συμβούλιο και την Επιτροπή αλλά και την Κίνα. Εδώ εσεί είστε ο κύριο ομιλητή. Ήρθετε από πολύ μακριά για να μας μιλήσετε. Οι λοιποί ομιλητές δεν θα έχουν τόσο χρόνο στη διάθεσή τους. Γι' αυτό και θα σας παρακαλέσω, αγαπητοί συνάδελφοι, να είσαστε όλοι πολύ σύντομοι. Κύριε Κίλγραμ, λυπούμε που δεν μπορώ να σας διαθέσω τόσο χρόνο ομιλίας. Πέντε με επτά λεπτά μόνο, αλλά σας καλωσορίζω σας γνωρίζω ήδη, έχουμε συναντηθεί στην Φιλανδία. Είστε δικηγόρος που ασχολείται με τα θέματα του διεθνούς δικαίου και έχετε συντάξει ή συμμετάσχει μάλλον στη σύνταξη της μελέτης για την Φόν Γκόγκ. Και επίσης ε, έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα και μελετήσει το φαινόμενο των, ε, του παράνομου εμπορίου ε, οργάνων του ανθρώπου για μεταμοσχεύσει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ασφαλώς μπορείτε να λάβετε, αν σας ενδιαφέρει, ε, το κείμενό μου το οποίο έχω ήδη διαθέσει στην είσοδο και παρακαλώ να με διακόψετε, Πρόεδρε, όποτε θεωρείτε ότι έχω ξεπεράσει τον χρόνο μου. Έρχομαι λοιπόν εδώ να μιλήσω για τα θέματα των, ε, πιστών της ομάδας Falun στην Κίνα άλλος ένας Γκάο, Γκάο που δεν είναι συγγενής ε, του εδώ κυρίου Γκάο, δίνει αντίστοιχε ε, μαρτυρίες. Ο Γκάο Σισέν ε, ήταν ένας από τους μεγάλους δικηγόρους που αγωνίστηκαν για να περασπιστούν την, το κίνημα Falun Έχει φυλακιστεί, δεν ακούστηκε καν από, την, από το δικαστήριο η επιχειρηματολογία του. Απευθύνθηκε όμως αυτός στην ομάδα των στην Διεθνή Ομάδα Ειδικών ε, φυλακίστηκε, βασανίστηκε για πέντε εβδομάδες, πέντε φρικτές εβδομάδες. Τώρα είναι άγνωστο το που κρατείτε δεν έχει διεθνής αμνηστία πληροφορίες. Επίσης ε, η γυναίκα του και η κόρη του υπέστησαν σημαντικές ε, παρενοχλήσεις σε όλη αυτή την περίοδο. μα είπαν ότι έχει περάσει πολύ ε, σε πολύ σκληρές συνθήκες, ε, χωρίς ε, επαρκή τροφή, νερό, θέρμανση. Δεν είναι γνωστό το που κρατείτε. Και πρέπει να σας πω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ε, στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας που δημιουργήθηκαν ε, την εποχή του ΜΑΟ με βάση τα παραδείγματα του Στάλιν και του Χίτλερ και του Τρίτου Ράιχ και που επιτρέπουν στο καθεστώς της Κίνας για τέσσερα χρόνια τουλάχιστον ε, να ε, κρατούν κάποιον χωρίς να υπάρχει κανένας ε, τρόπος, κανένα δικαίωμα προσφυγής, παρέμβασης, αντίδρασης ή έφεσης. Και μάλιστα από αυτά παράγονται και προϊόντα τα οποία έρχονται στη Δύση, Χριστουγεννιάτικα, Στολίδια και άλλα. Έχουμε εδώ να κάνουμε με ένα καθεστώς ολοκληρωτικό που επιτρέπεται στο οποίο επιτρέπεται ε, κάθε παρέα βίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χάρη στην πολιτική της Δύσης. Βλέπετε εδώ και τη φωτογραφία της ε, ακολούθου της Φάλων Γκόγκ η οποία ενώ πριν ήταν επαγγελματίας και μάλιστα και εραστέχνης ηθοποιός, συνελήφθη, βασανίστηκε και δεν θα σας διαβάσω τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της ζωής της γιατί ε, είναι πραγματικά πολύ τραγικές. Βλέπετε λοιπόν ότι συνεχίζονται οι διώξει εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον ει βάρο των ανθρώπων αυτών. Εγώ αγαπώ ιδιαίτερα την Κίνα και είμαι πολύ περήφανο για, την, ε, για τη χώρα αυτή. Όμως ε, ξέρουμε, πολύ, ε, ξέρουμε ότι είναι οι παραβιάσεις των ανθρωπινών δικαιωμάτων ε, συνεχείς και εκτεταμένες. Υπάρχουν πολλές αναφορές ότι μέλη της Φαλον Κόγκο, εκτός του ότι βασανίστηκαν, κρατήθηκαν παράνομα, έχουν ακόμη και εκτελεστεί προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα όργανα τους για μεταμοσχεύσεις, για το εμπόριο των μεταμοσχεύσεων. Ξέρετε ότι πρόκειται για μια οργάνωση η οποία ασχολείται μόνο με τον διαλογισμό, δεν έχει καθόλου βίαιη συμπεριφορά οι πρακτικές τα υπόλοιπα τα βλέπετε μέσα στην έκθεσή μου. Το 92 ξεκινήσανε και μέχρι το 99 ήταν τόσο ισχυρή, ισχυρό το κίνημα που, θυμ, που ανησύχησε το καθεστώ τη Κίνα για την επέκταση τη δυναμή του. Συνεχίζουν λοιπόν από... Μάλιστα με τις, με τις εκτιμήσεις ε, της κυβέρνησης ε, από μηδενικά νούμερα περίπου το 92 μέχρι το 99 είχαν φτάσει σε αρκετά εκατομμύρια, σε πολλές δεκάδες εκατομμυρίων ε, το 1999 έως και 70 έως 100 εκατομμύρια. Πολλοί εκλήθησαν ε, από τις αρχές ε, να παρετηθούν, να εγκαταλείψουν το κίνημα, συνελήφθησαν, βασανίστηκαν και όταν ακόμη δεν δήλωσαν με τα πολλές φορές εξαφανίστηκαν σε συνθήκες κράτησης και ε, δολοφονήθηκαν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα όργανα τους και μετανοσμοσχεύσεις οι οποίες σε κύριο αποδέκτη έχουν δυτικούς τουριστές. Προχωρώ πολύ γρήγορα για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Θα ήθελα απλώ να πω ότι μόνο οι ακόλουθες φαλούν Gong στα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας και τις φυλακές υποβάλλονται σε συστηματικούς ελέγχους ε, είτε σωματικής κατάστασης, είτε φυσικής κατάστασης, είτε αιματολογικούς, που είναι απαραίτητο βέβαια για να επαληθευθεί ότι είναι χρήσιμα τα όργανα τους για τις μεταμοσχεύσεις. Η, αρχή η φρικτή αυτή αρχή που ακολουθούν είναι ότι αν υπάρχει μεταξύ αυτού εδώ του προσώπου που βλέπετε ε, και βρίσκεται σε ένα στρατόπεδο κρατήσεω και κάποιου που έρχεται από το Ελσίνκι για να πάρει ένα όργανο για μεταμόσχευση και μπαίνει μέσα σε ένα, σε ένα ε, νοσοκομείο τη Σανκάη, αυτή την κυρία θα την πάρουν από το στρατόπεδο. Ε, όπου κρατείται από το στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας μόνο και μόνο με αυτό το κριτήριο τη συμβατότητα δηλαδή, θα την εκτελέσουν και θα πάρουν όλα τα όργανα προκειμένου να σα τα μεταμοσχεύσουν, να σα μεταμοσχεύσουν εσά το σηκώτη που ενδεχομένω χρειάζεστε. Αυτή είναι η αποτρόπαιη κατάσταση που έχουμε στην ε, Κίνα. Δεν υπάρχουν ε, ε επαρκείς ε, πόροι μεταμοσχεύσεων από κρατουμένους θανατοποινίτες που εκτελέστηκαν και μετά αξιοποιήθηκαν τα όργανά τους ώστε να δικαιολογείται ο αριθμός, ο τεράστιος αριθμός των μεταμοσχεύσεων που λαμβάνουν χώρα στην Κίνα. Δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα ε, δωρεάς οργάνων, δεν υπάρχει καν ε, η κουλτούρα, η νοοτροπία του, της διάθεσης των οργάνων ε, ενός νεκρού από την οικογένειά του. Το μόνο φαινόμενο που μπορεί να εξηγήσει τους τόσους μεγάλους αριθμούς μεταμοσχεύσεων είναι αυτές ακριβώς οι εκτελέσεις των μελών το, ε, του κινήματος Φαλούν Γκόγκ. Πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι από από τις ε, ε, από τα, τηλέφω, από τα νοσοκομεία της Κίνας μας δίνουν πληροφορίες για τέτοιου είδους εκτελέσεις. Μέχρι και 41.500 νεκρούς νομίζω ότι έχουμε θρηνήσει ακριβώς για να χρησιμοποιηθούν τα όργανα τους. Αλλά θα δείτε τις λεπτομέρειες στην έκθεση. Υπάρχουν ε, πολυάριθμες καταδίκες για ορισμένους οι οποίοι ε, έχουν ε, κατηγορηθεί για πολλά αδικήματα, ενώ τα μέλη της Falun βρίσκονται κρατούμενοι χωρίς καν να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, να έχουν διαπράξει το παραμικρό έγκλημα. Στα στρατόπεδα αυτά καταναγκαστικών έργων, στα κάτεργα αυτά, είναι δεκάδες χιλιάδων ε, αυτοί που κρατούνται από τη Falun και που εκτελούνται. Έτσι λοιπόν, ε, για να προχωρήσω λίγο πιο γρήγορα ακόμη, μια δυνατότητα που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε νομικά θα ήταν να εφαρμοστεί η λεγόμενη εξοεδαφική ε, νομοθεσία, δηλαδή ένας Καναδός ο οποίος θα έρθει από τον Καναδά για να πάει στην Κίνα να ε, δεχθεί μεταμόσχευση οργάνων ανθρώπου που έχει παράνομα εκτελεστεί, θα ήταν υπόλογος με βάση το καναδικό δίκαιο όταν επέστρεφε στη χώρα του. Αλλά ταυτόχρονα πιστεύω ότι θα πρέπει να απαγορευτεί ε, με οποιονδήποτε τρόπο στις ευνομούμενες χώρες της Δύσης η χρήση τέτοιου είδους οργάνων. και κάθε δείγμα που έχουμε και σε σχέση με τη Φαλούν Κόγκα αλλά και με όλα τα υπόλοιπα ανθρώπινα δικαιώματα μας υποδεικνύει ότι πρέπει οι λοιπές κυβερνήσεις του κόσμου να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικές έναντι της κυβέρνησης της Κίνας, έναντι του καθεστώτος, σε οποιοδήποτε συναλλαγή για να πιεστεί να επιστρέψει στις τάξεις των κρατών που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ο λαός της Κίνας, τον οποίο σέβαμε και αγαπώ πολύ, έχει αρετές, μοναδικές, εγκαρτέρησης, υπομονής και αγαθότητας και πιστεύω ότι έχει τη θέση του μέσα στη διεθνή κοινότητα. Η Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κιλγκόρ. Είναι πίστευτο πραγματικά ότι μια φιλιρινική ομάδα, ε, ε, κοινότητα ανθρώπων όπως οι οπαδοί του Falun μπορούν να γίνονται αντικείμενο τέτοιας εκμετάλλευσης. Θα ήθελα να ε, ακούσουμε τώρα την εκπρόσωπο του Ινστιτούτου της Βιέννης. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα να συμβάλλω στην σημερινή συζήτηση. Μου ζητήθηκε να μιλήσω για θέματα πολιτικής της ε, Ευρώπης απέναντι στην Κίνα για θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων. Έχουμε στοιχεία από 60 εμπιστευτικές ε, συνεντεύξεις και άλλη έρευνα που έκανα τα τελευταία δύο χρόνια. Θα σας παρουσιάσω τις προσωπικές μου βέβαια απόψεις, χωρίς αυτές να απηχούν τις απόψεις κανενός οργανισμού. Έθεσα ορισμένα ερωτήματα. Λειτουργεί ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Κίνα. Δεύτερον, υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις. Και τρία, πού μπορεί η Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πορευτούν από εδώ και πέρα. Για το πρώτο ερώτημα, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει, έχει δηλώσει κατά επανάληψη ότι ο διάλογος έχει νόημα εάν υπάρχει αρκετή πρόοδος επιτόπου. Όπως έχω ξαναπεί, ο διάλογος για πρώτη φορά αξιολογήθηκε από εξωτερικό εμπειρογνώμονα φέτος. Ωστόσο, η αξιολόγηση αυτή εντοπίστηκε μόνο στο πώς μπορεί να βελτιωθεί ο διάλογος και όχι εάν αξίζει να συνεχιστεί. Αρνητική αξιολόγηση του διαλόγου είχε νόημα να αποφευθεί, διότι οι χώρες μέλη δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε άλλη εναλλακτική πολιτική. Ο διάλογος βοηθεί να προληφθεί η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα ψήφισμα των ΗΠΑ. Δεύτερον, πρέπει να βασίζεται ε, σε αμοιβαίο σεβασμό και να μην αναφέρεται σε κανένα, και δεν αναφέρεται σε κανένα από τις ουσιώδεις ανησυχίες. Ο διάλογος γίνεται ανάμεσα σε ένα μικρό αριθμό αξιωματούχων. Είναι περίπλοκες οι μεταρρυθμίσει, ο στόχος είναι πολύ φιλόδοξος, αλλά να ισχυριζόμαστε τώρα ότι τέτοιο διάλογος μπορεί να λειτουργήσει σαν δούριο ύπος, αυτό πραγματικά δεν πείθη κανένα. Τον Φεβρουάριο του 2000, ο τότε Επίτροπος Κρίστοφερ Πάτεν είχε σχολιάσει ως εξή στο Κοινοβούλιο, μάλιστα, τον διάλογο αυτό. πρέπει να μπορούμε να σας πείσουμε ότι ο διάλογος αυτός οδηγεί κάπου. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είχε πει τότε, είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε τις επόμενες εβδομάδες. Σχεδόν 10 χρόνια μετά εξακολουθεί η πρόκληση αυτή να υπάρχει. Η Κίνα γνωρίζει τώρα ότι η Ευρώπη δεν πρόκειται να επιστρέψει, επιστρέψει στα ψηφίσματα αυτά ακόμα και αν δεν λειτουργήσει ο διάλογος. Προσπάθησε η Κίνα να πείσει την ε, Ευρώπη ότι αξίζει ο διάλογος. Και κάθε Προεδρία έχει κάνει και μία μικρή παραχώρηση για να δικαιολογηθεί η ύπαρξη του διαλόγου. Παραδείγματα. Στον διάλογο τον Οκτώβριο του 1999 υπό Φιλανδική Προεδρία ανακοινώθηκε ότι η Κίνα επρόκειτο σχεδίαζε να καταργήσει θανατική ποινή. Είχε θεωρηθεί τότε αυτό σημαντικό βήμα προόδου στον διάλογο και αναμένονταν αποφάσεις. Αργότερα κατάλαβαν οι αξιωματούχοι ότι η ανακοίνωση αυτή δεν ήταν παρά μια διπλωματική κίνηση για να συγγύσουν οι κριτικές σχετικά με την αναποτελεσματικότητα του διαλόγου. Μετά από πολλά χρόνια διαπραγματεύσεων, εν τέλει επετράπησε έναν ε, ειδικό απεσταλμένο να, εξετάσει, να μεταβεί στην Κίνα για να εξετάσει θέματα βασανιστήριων. Αυτό θεωρήθηκε ότι ήταν ιδιαίτερη χάρη που έκαναν οι Κινέζοι στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι ήταν Ευρωπαίος ο παρατηρητής αυτός. Διακόπτη πρόοδος μπορείτε παρακαλώ να ε, μιλείτε λίγο πιο αργά για να σας προλαβαίνουν και μεταφραστές. Συνεχίζω λοιπόν, το 2005 προσκλήθηκε το πρόσωπο αυτό και ε, όπως είπα θεωρήθηκε ότι ήταν μια μεγάλη χάρη που έκαναν οι Κινέζοι, ειδικά στους Ευρωπαίους επειδή ήταν Ευρωπαίος αυτός ο παρατηρητής. Επέμειναν οι Ευρωπαίοι ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα του διαλόγου, αλλά αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό και ιδιαίτερα διότι ήταν και όρος τον οποίο είχε θέσει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για να ξαναρχίσει τον διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την Κίνα. Στην ομάδα διακυβερνητικού συντονισμού για όλους τους διαλόγους με την Κίνα, που την ε, γνωρίζουμε ως η διαδικασία της Βέρνης, φάνηκε καθαρά ότι σε όλους τους, συνομιλητές, σε όλους τους συνομιλητές της η Κίνα είχε κάνει αυτήν την χάρη, την ίδια και μοναδική. Άρα αυτά δεν οδηγούν σε πολλά πράγματα και ούτω ή άλλω η αλλω η ευρωπη δεν ε, χαίρει πλέον ε, τέτοια ειδική μεταχείριση μεταχείρισης από τους Κινέζους. Τώρα, μεταξύ 2004 και 2006 εκδόθηκαν ε, πλήρωνε ανακοινώσει από το Συμβούλιο των Υπουργών που εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόλυση από τις φυλακές διαφόρων προσώπων όπου είχε θέσει τις υποθέσεις τους υπόψη των Κινέζων. Εγώ δεν έχω δει ούτε έναν αξιωματούχο της Ένωσης που να προσπαθήσει καν να μην πείσει ότι κάποιο ρόλο έπαιξε η Ευρώπη στην, απο... στην απόλυση των προσώπων αυτών. Πάντα ήταν μετά από πίεση των Αμερικανών. Ίσως τώρα ο διάλογος αυτός να βοηθεί να βελτιώνονται οι συνθήκες κράτησης ορισμένων κρατουμένων. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ένωση, από όσο ξέρω εγώ τουλάχιστον, δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η ίδια επέτυχε την απόλυση ιουδήποτε κρατουμένου ή υπερασπιστού ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στην Κίνα την τελευταία δεκαετία. Στην πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο να διαπιστώσει κανείς ποια είναι ε, η επίδραση του διαλόγου στην Κίνα. Ασφαλώς, πολύ σημαντικότερο ρόλο παίζουν εσωτερικοί παράγοντες. Και ο διάλογος αυτός δεν είναι ούτε επαρκής, ούτε αναγκαία συνθήκη για την λήψη οποιασδήποτε απόφασης από πλευράς των Κινέζων. Προσωπικά θεωρώ ότι η ε, επίδρασή του είναι μάλλον απίθανη. Ένα άλλο στοιχείο που σημειώνω είναι ότι οι περισσότεροι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο διάλογο με τους Κινέζους δεν γνωρίζουν την κινέζικη γλώσσα. Δεν μπορούν καν να παρακολουθήσουν ε, σημαντικά θέματα που ε, συμβαίνουν στην Κίνα. Ο ο ρόλο του σεμιναρίου είναι να επηρεαστούν οι συζητήσει αυτέ. Μα πώ είναι δυνατόν να επηρεαστούν, αν δεν γνωρίζει κανεί τι λεπτομέρειε των συζητήσεων αυτών. Στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γίνεται περιοδική επανεξέταση, έγινε και τελευταία τον Φεβρουάριο και μετά από μία δεκαετία και κλεισμένων των θυρών, τούτη εδώ που ήταν και δημόσια η συνεδρίαση δεν απαιτέλεσε καμία ιδιαίτερη πρόκληση. Όλοι συνέκριναν στον ίδιο στόχο της κριτικής. Οι δηλώσεις που, έκαναν που έγιναν από χώρες ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέδειξαν την ευρωπαϊκή ποικιλότητα. Ούτε μία σύσταση δεν έγινε από όλους τους Ευρωπαίους αγορητές στη διάρκεια της ε, διοργάνωσης αυτής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την τάση να θέτει πάρα πολλά θέματα ταυτόχρονα. Το 2001 το Συμβούλιο έθεσε μια ε, ατζέντα. Το 2003 είπε ότι θα άρει τον, ε, το εμπάργο όπλων μετά από την ε, συμφωνία που είχε επιτευχθεί με, που όπου ζητούσε απόλυση των κατουμένων της Τέναν ελευθερία έκφραση γνώμης και άλλα θέματα, τα οποία έχουν επαναληφθεί ξανά και ξανά, αλλά συνδέονται μοναχά ως υποπαράγραφος με την άρση του εμπάργου των όπλων. Μόνο όταν οι, ε, μετά όμως οι Ηνωμένε Πολιτείες παρενέβησαν και πίεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην άρει το εμπάργο των όπλων. Όταν αντιλήφθησαν πλέον οι Κινέζοι ότι ε, ε, δεν θα ήρετο ο αποκλεισμό, το εμπάργο όπλων, έτσι έστω και αν έκαναν τις παραχωρήσει που ζητούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε γιατί να τι κάνουν. Τώρα έχει έχουν περιθωριοποιηθεί οι διμερείς συζητήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το μήνυμα είναι, τελικά που δίνει η Ευρώπη, είναι ότι ενδιαφερόμαστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά όχι και τόσο πολύ. Μέχρι τώρα λοιπόν ο διάλογος δεν έχει επιτύχει ως μηχανισμός να καταλήξει στο να δοθούν κοινέ συστάσεις και έχουν μείνει εκτός του επισήμου διαλόγου οι εκπρόσωποι των μη κρατικών οργανώσεων. Για την επανάληψη του διαλόγου το 1997 είχε λεχθεί ότι επρόκειτο να ανοιχθεί ο διάλογος και σε εκπροσώπους των μη κρατικών οργανώσεων. Και ανοίχθηκε πράγματι. Αλλά μετά επειδή, επειδή απαγορεύτηκε το China Democracy Party και οι μη κρατικέ οργανώσεις απεχώρησαν. Κάποιο διάστημα αργότερα απεφάσισαν να επανέλθουν, αλλά δεν τους επετράπη. Τελειώνοντας, Πού μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να οδεύσουν από εδώ και πέρα. Εγώ θεωρώ ότι έχει έρθει η ώρα να επανεγκύψετε στην πολιτική απέναντι στην Κίνα. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ξανά και ξανά συστάσεις για την ενίσχυση του διαλόγου. Ακούμε διαρκώς τα ίδια μηνύματα. Στο παρελθόν η προσέγγιση αυτή δεν απέδωσε αποτελέσματα, διότι είναι βολικό όχι μόνο για τους ηγέτες της Κίνας, αλλά και για τους ηγέτες της Ευρώπης να διατηρούν τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα δεύτερο, δευτερεύον επίπεδο. Στο περιθώριο. Για να μεταφέρει το μήνυμα της ανησυχίας και για να ζητήσει απάντηση σε συγκεκριμένε υποθέσεις, ατομικές υποθέσεις, δεν χρειάζεται τον διάλογο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να τα κάνει αυτά μέσω, μέσα άλλων οδών της διπλωματικής οδού ή και σε άλλους διαλόγους, σε διμερείς διαλόγους. Εάν ζητεί η Ευρώπη, αν επιζητεί κάποια αποτελέσματα, θα πρέπει να θέσει ένα θέμα κάθε φορά. Για παράδειγμα, την αναστολή των θανατικών εκτελέσεων. Αυτό θα ήταν μια ρεαλιστική προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε μάλιστα να δεχθεί να διακοπεί ο διάλογος εάν η Κίνα αποφασίσει να κάνει την παραχώρηση που τη ζητείται στο ένα σημαντικό αυτό θέμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει κατ' επανάληψη, κοιμάστε και την τελευταία εβδομάδα ακόμη, να μπει στι συμφωνίε μια ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ συμφωνώ, αλλά τι θα σημάνει η ρήτρα αυτή. Εγώ θα συμβουλεύσω την υποεπιτροπή σας να καταθέσει ένα σχέδιο ψηφίσματος για να αναλάβει τη δέσμευση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δέχεται συμφωνίες με χώρες που έχουν κυρώσει την ICCPR. Αυτό μπορεί να αποδώσει. Από εδώ και πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει και κυρώσει συνθήκες με χώρες που δεν έχουν κυρώσει την ICCPR όπως το, το Πακιστάν. Μέχρι τώρα όμως δεν έχει, αν δεν κάνω λάθος, καμία συμφωνία συνεργασία. Ιδεοδό όλε οι συμφωνίε με τρίτε χώρε θα έπρεπε να υπόκεινται στον όρο αυτό, τη κύρωση τη ICCPR. Και ελπίζω ένα τέτοιο ψήφισμα, εάν ενδεχομένω το καταθέσετε, να μην αφήσει απ' έξω την Κίνα. Ώστε επιτέλου να παρακινηθεί η χώρα αυτή να ακυρώσει την ICCPR. Πιστεύω ότι αυτό θα ήταν ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε για την πολύ ψύχρεμη αυτή η ανάλυση του διαλόγου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Πιστεύω την ε, σύσταση αυτή ότι θα πρέπει το SCPR να γίνει δεκτός ε, προδιαγραφή δασική, θα πρέπει να την διατηρήσουμε πιστεύω όλοι, να την έχουμε όλοι υπόψη και μίλησε μόνο ότι σήμερα τίφτε σε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνα, η οποία δίνει και πολύ περισσότερες εξουσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ω προ τι ε, συμφωνίες. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή. Τον κύριο Μπρατ Άνταμς, ε, συγγνώμη, τον κύριο Σάμπας, διευθυντή του Ιρλανδικού Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπου διεξάγονται και τα σεμινάρια εν ώψη του επίσημου διαλόγου. Πρόκειται για σεμινάρια τα οποία ξέρουμε πως έχουν χρησιμοποιηθεί ως πρόφαση, ως δικαιολογία, ώστε να υποβαθμιστεί η σημασία των ε, θεμάτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διαλόγου αυτού. Κύριε Σάμπας. Είναι εύστοχη αυτή η παρατήρηση, κύριε Σέβα. Εγώ, Πρόεδρε, δεν έχω συμμετάσχει ενεργά στον πολιτικό διάλογο και σε δεν είμαι σε θέση να απαντήσω στην ερώτησή σα ω προ τι ε, ε, επιπτώσεις, των, ε, την αντανάκλαση αυτών των σεμιναρίων σε άλλε διαδικασίε. Απλώ. θα ήθελα να σα επισημάνω ότι αυτά τα σεμινάρια λαμβάνουν χώρα εδώ και δέκα χρόνια περίπου. Έχει ξεκινήσει ο, ο διάλογος από τα τέλη τη δεκαετία του 90 Έχω συμμετάσχει σε αυτά και πολλές φορές έχω διοργανώσει από πλευράς της, Ευρωπα... Ευρώπης τα σεμινάρια αυτά. Τα βλέπω λοιπόν να εξελίσσονται στον χρόνο. Είναι διαδικασίες επώδυνες, δύσκολες ασφαλώς όπως αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι από τους εδώ παρισταμένους. Πρόκειται περισσότερο για εργαστήρια στα οποία συμμετέχουν ε, επιστήμονες ε, από τα πανεπιστήμια της Ευρώπης. μια αρκετά ευρεία εκπροσώπηση ευρύ φάσμα εκπροσώπηση, από κινέζικα πανεπιστήμια, όπου κατά καιρού είχαμε πιο ευρεία εκπροσώπηση, ενώ τώρα μάλλον βλέπουμε να περιορίζεται το πεδίο ε, των ε, ερευνητικών κέντρων και ιστοτών που μας αποστέλουν επιστήμονες. Τώρα πια έχουμε μόνο από το Πεκίνο και περιοριζόμενους και από εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ακόμη εκπροσώπους και της Διεθνούς Αμνηστίας και του Human Rights Watch όπως και άλλων, ε, άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ήταν δύσκολε λοιπόν οι συνθήκε υπό τι οποίε οργανώσαμε τα σεμινάρια τελευταία χρόνια. Ένα από αυτά μάλιστα δεν έλαβε καν χώρα. Ένα άλλο τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά τελευταία στιγμή ε, την ώρα που ήταν ε, ήδη καθισμένοι στα τραπέζια και ξεκίνησαν τις συζητήσεις τους ε, οι συμμετέχοντες, ματαιώθηκε. Στο Galway, το κέντρο μας στην Ιρλανδία, ανέλαβε, πιστεύω, με επιτυχία τη διοργάνωση των σεμιναρίων, δύο από αυτών, που ήταν δύσκολο, όπως σας είπα, στην διοργάνωσή τους, αλλά και επίσης πολλές φορές προβληματική επιλογή των θεμάτων, όπως και των ε, συμμετεχόντων. Για δε τους συμμετέχοντες, επιτρέψτε μου να πω, ξεκινώντας ότι έστω και με ευρία συμμετοχή των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων και των εκπροσώπων και από τη Human Rights Watch και τη Διεθνή Αμνηστία τελευταία φορά που σας εξήγησα νωρίτερα, λίγοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι αποτελούν ε, persona non για την κινέζικη κυβέρνηση, για το, κοινωνικό, για το κινέζικο καθεστώς. Και βέβαια όταν πρόκειται να πάμε στο Πεκίνο, στην Κίνα για να γίνει το σεμινάριο εκεί, προφανώς τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ. Θα πρέπει να σας πω ότι δεν κάνω παρασκηνιακές συμφωνίες ε, εγώ με το καθεστώς της Κίνας προκειμένου να επιλεγεί ο ένας ή ο άλλος ε, επιστήμονας. Πρόκειται για ανοιχτή αντιπαράθεση ε, και πρέπει να πω επίση ότι η δική μα πλευρά, η ευρωπαϊκή πλευρά, δεν έχει έλεγχο στο ποιο επιλέγεται από το κινέζικο καθεστώ. Με τα τελευταία λοιπόν σεμινάρια ε, αγγίξαμε μια σειρά θεμάτων, ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα σε πολλέ του πτυχέ, χωρί ε, ταμπού, τη συζήτηση παραδείγματι τη θεραπευτική ποινή ε, ή των κατέργων ή του δεδικασμένου ή των βασανιστήριων, συνθήκες κράτησης. Ασφαλώς θα αντιλαμβάνεστε και ότι για ορισμένα θέματα είναι αδυνατό να συμφωνήσουμε με τους Κινέζους για τη συμπερίληψή τους ε, στην ημερήσια διάταξη, όπως για παραδείγματι το θέμα το οποίο συζητήθηκε νωρίτερα για την Falun είναι ένα θέμα το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα απέρριπταν ω αντικείμενο συζήτηση Κινέζοι. Εγώ προφανώ δεν θα ήθελα καν να είμαι μέσα στην αίθουσα την ώρα που θα διατυπωνόταν η πρόταση για συμπερίληψη τη ημερήσια διάταξη ενό σεμιναρίου. Αυτέ είναι οι πραγματικότητε τι οποίε αντιμετωπίζουμε στην οργάνωση των σεμιναρίων. Και εδώ εγώ θα ήθελα να πω ότι το καλύτερο μερικέ φορέ είναι και ο εχθρό του καλού. Επιτρέψτε μου να σημειώσω, γιατί δεν ε, περίμενε ερχόμενο εδώ ότι θα ακούσω τέτοιε ε, συγκεκριμένες και ε, ε, συγκεκριμένε τοποθετήσει και μάλιστα τοποθετήσεις οι οποίες τρέφονται κατά της ακαιρεότητα και του επιστημονικού χαρακτήρα των σεμιναρίων αυτών, δεν θέλω να πω ότι δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι δεν έχει επιτευχθεί τίποτα στη διαδικασία αυτή. Όπως επίσης είναι πολύ σκληρό το να ισχυρίζεται κανείς ότι ε, μόνο μία ε, ότι έχουμε μόνο θετική, θετικό αντίκτυπο, ότι έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα. Κανεί δεν ισχυρίζεται ότι μπορεί να το επιτύχει αυτό ένα σεμινάριο, ούτε εδώ, ούτε στην Ευρώπη ολόκληρη. Έχουμε τέτοιε ψευδεστήσει. Και δεν θέλω παρακαλώ τα λόγια μου να ερμηνευθούν ω ε, αμφισβήτηση των ισχυρισμών των άλλων ομιλητών για τα προβλήματα στην Κίνα. Αλλά το να λέει κανεί ότι δεν, δεν έχει υπάρξει καμία θετική εξέλιξη, καμία βελτίωση, πάλι μου φαίνεται άδικη εκτίμηση. Τα θέματα αυτά, τα οποία γνωρίζω εγώ καλύτερα από όλους, αφού είναι ε, η ειδικότητά μου η επιστημονική και έχω συμμετάσχει σε ακαδημαϊκά σεμινάρια και άλλες δραστηριότητες που προχωρούν εκ παραλίλου και πολλές φορές χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κυρίως θέματα θανατικής ποινής. Εδώ και μια δεκαετία περίπου που ασχολούμαι με το θέμα αυτό και την Κίνα, βλέπω σημαντικές ε, αλλαγές, όπως σε παραδείγματι την ε, αυτεπάγγελτη προσφυγή στο Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο ή Δικαστήριο του Λαού της Κίνας. Ε, πολλές είναι οι εξελίξεις ε, που βλέπουμε, πολλές οι βελτιώσεις. Δεν είναι ασήμαντες. Επίσης έχει βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα του διαλόγου γιατί εδώ πάλι οι επιστήμονες βλέπουν ε, την ε, αλλαγή περισσότερο πιο καθαρά από τι άλλοι. Εμείς ζητούμε με άλλους επιστήμονες και βλέπουμε πώς αλλάζει δική τους συμπεριφορά και στάση. Τα τελευταία δέκα χρόνια είναι αισθητή η εξέλιξη. Κυρία Κίντσελμπαχ είπε νωρίτερα ότι είχαν ισχυριστεί οι Κινέζοι σε κάποια συνεδρία ότι ήταν έτοιμοι να καταργήσουν τη θανατική ποινή δεν το θυμόμαι εγώ αυτό, δεν ε, νομίζω ότι είπαν πως είναι έτοιμοι να καταργήσουν τη θανατική ποινή. Μάλλον θα είπαν ότι μακροπρόθεσμα στοχεύουν στην κατάργηση θανατικής ποινής και ότι βράχει πρόθεσμα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα όπως τα αντιμετωπίζουν. Πάντω, θα ήθελα να σημειώσω ότι γενικά βλέπω μια βελτίωση. Πριν από 10 χρόνια που ξεκίνησα με το θέμα αυτό, επέμεναν πολύ οι Κινέζοι, δεν υπήρχε καμιά ευελιξία προς θανατική ποινή. Ε, μας έλεγαν οι αρχές, οι εκπροσωποί τους ότι ε, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο βρίσκει σύμφωνο τον Κινέζικο λαό, ότι ο Κινέζικος λαός εκ είναι υπέρ της θανατικής ποινής και ότι μόνο τους Ευρωπαίους ενοχλεί θανατική ποινή. Και όμως εδώ βλέπουμε αλλαγές. Βλέπουμε μια συνολική αλλαγή στάση. Βλέπουμε ότι ο στόχο στόχος μακροπρόθεσμα ορίζεται και νομίζω ότι υπόθηκε αυτό από κάποιον εκπρόσωπο επίσημο τη κυβέρνηση σε ένα Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μακροπρόθεσμο στόχο λοιπόν είναι η κατάργηση τη θανατική ποινή. Επίση καταργείται η θανατική ποινή, περιορίζεται ε, και έτσι δεν, δεν επιβάλλεται πλέον για εγκλήματα οικονομικού χαρακτήρα ή μη βία εγκλήματα. Είναι μια πρόοδο αυτό. Πιστεύω ότι ναι, είναι αναμφίβολα μια πρόοδο αυτό. Τώρα, εάν η πρόοδος ε, σημειώνεται λόγω της δικής μας παρέμβασης, δεν ξέρω. Πάντως δεν νομίζω ότι, απο, ότι προκύπτει ως απόρρια των πιέσεων των Αμερικανών, γιατί οι Αμερικανοί δεν γνωρίζω ποτέ να πίεσαν τους Κινέζους για κατάρριση εναντικής ποινής. Θα συμφωνήσω όμως, ελπίζω μαζί μου, να ε, στο ότι φυσικά δεν μπορούμε εμείς να διεκδικήσουμε τα ε, εύσημα ε, των βελτιώσεων αυτών, αλλά από την άλλη γιατί να μην δούμε ότι υπάρχουν οι βελτιώσεις, γιατί να αρνηθούμε ότι υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Το ότι υπάρχει ο διάλογος με όλες τις δυσκολίες, το ότι υπάρχει ανταλλαγή απόψεων, ούτε αιτία του προβλήματος είναι ενδεχομένως, ούτε και η μαγική σφαίρα, η πανάκια η οποία θα φέρει τη λύση κάποια μέρα. Είναι ένα λιθαράκι. Αλλά νομίζω πολύτιμο λιθαράκι. Εξάλλου, οι επιστήμονε είναι και κομμάτι τη κοινωνία των πολιτών. Στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ένα τομέα θα έλεγα ειδικό σχετικά καινοτόμο, βλέπουμε ότι υπάρχουν νέε έδρε. Εγώ είμαι πρόεδρο αντίστοιχα τη έδρα μου στο Πανεπιστήμιό μου. Ε, Όπω και άλλοι συνάδελφοι αναλαμβάνουν ε, έδρε ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε, διάφορες, ε, διάφορα πανεπιστήμια, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και αγωνιζόμαστε όπως κάθε ε, πανεπιστημιακός ερευνητής να βελτιώνουμε τον τομέα που, ε, στον οποίο έχουμε αφοσιωθεί, αφοσιωθεί. και πιστεύω ότι το ίδιο κάνουν και οι επιστήμονες της Κίνας. Και προσπαθούν να βελτιώσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα τους. <coughs> τα σεμινάρια αυτά προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για ε, γνωριμία και δεσμούς, ανάπτυξη δεσμών μεταξύ Ευρωπαίων και Κινέζων επιστημόνων αποτελούν ένα πεδίο ανταλλαγή απόψεων ανθρώπων που βρίσκονται στον πανεπιστημιακό χώρο που αγωνίζονται και ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολλά είναι τα θέματα στα οποία προσπαθούμε να βελτιώσουμε, βλέπουμε ελλείψεις και θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των ε, σεμιναρίων μα. Θα το επιτύχουμε πιστεύω, Συνεχίζουμε την προσπάθεια, αλλά παρακαλώ και εσεί αναγνωρίστε την θετική συμβολή αυτών των σεμιναρίων όλα αυτά τα χρόνια ως προς το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Ευχαριστώ πολύ, καθηγητά κύριε Σάμπας. Ασφαλώς είναι πολύ χρήσιμο να υπάρχει αυτός ο διάλογος. Μίλησατε για διάφορα βήματα που θα πρέπει να ε, πραγματοποιηθούν ακόμη. και εμείς ε, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελπίζουμε να γίνει κύρωση ενός κεντρικού νομοθετήματος που θα καλύπτει τα θέματα των δικαιωμάτων. Και τώρα θα παρακαλέσω τον κύριο Brad Adams, διευθυντή ε, του τομέα της Ασίας της Human Rights Watch, η οποία έχει δημοσιεύσει μια έκθεση για τις μαύρες φυλακές της Κίνας. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε να σας μιλήσω σήμερα. Τίποτα δεν θα ευχαριστήσει περισσότερο την κινέζικη κυβέρνηση παρά να ε, δει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μαλώνει για το πώς θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη τα θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Κίνα. Αυτά που είπε η Κάτριν ήταν πραγματικά έξοχα. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια ρεαλιστική άποψη για το τι πετυχαίνει ο διάλογος. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι και το ουσιώδες αυτό. Δεν θα πρέπει να καταναλώσετε πολύ χρόνο σε αυτό. Α μην ξεγελιόμαστε μόνο ότι ο διάλογο ή τα σεμινάρια έχουν οποιοδήποτε αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα. Δεν έχουν. Το ζήτημα είναι θα πρέπει να συνεχιστεί το σεμινάριο και ο διάλογο. Αλλά επειδή υπάρχουν όλα αυτά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κινέζικος λαό και η Κίνα, δεν πρέπει εδώ να μαλώνετε εσεί με, με τους δικούς σας, με του εαυτού σα, γιατί αυτό είναι αυτό που εξυπηρετεί την κινέζικη ηγεσία στην ουσία. Θα σας πω λίγα λόγια για ορισμένα πράγματα. Ε, αυτή είναι η έκθεσή μας για τις λεγόμενες μαύρες φυλακές που ανέφερε πριν ο πρέσβης. Έκθεση η οποία περιγράφει πώς ασκεί η κινέζικη κυβέρνηση μια πολιτική εξοδικαστικών κρατήσεων. Κλείνουν έναν από τους λίγους δρόμους που έχουν οι Κινέζοι, ο κινέζικος λαός να εκφράζει τα παραπονά του. Πριν από 20 χρόνια οι άνθρωποι στην Κίνα μιλώντας το βράδυ ή σε έναν ξένο στο δρόμο δεν θα τολμούσαν να ανοίξουν το στόμα τους. Αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει τώρα. Αν όμως προκαλέσετε μια αρχή, προκαλέσετε το κόμμα ή οργανώσετε κάποια αντίδραση, έχετε, ως κινέζο δηλαδή, ξεπεράσει τα εσκαμμένα. Έχετε υπερβεί τα εσκαμμένα. Δεν είναι ανεξάρτητα τα δικαστήρια, δεν υπάρχει ανεξάρτητη απονομή δικαιοσύνη. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν οι άνθρωποι είναι να, να πηγαίνουν τα παράπονά του όσο γίνεται πιο υψηλά, να τα φτάσουν δηλαδή στην ηγεσία του κόμματο, να πάνε στο Πεκίνο. Όμω οι αρχέ δεν θέλουν να φτάσει ο κόσμο στο Πεκίνο να πει στους αρμόδιους τα παράπονά τους. Έχουν λοιπόν ειδικού ανθρώπους που πάνε και βρίσκουν τους παραπονουμένους και τους επιστρέφουν στις ε, ιδιαίτερες πατρίδες τους. Τους συλλαμβάνουν, τους ε, εκφοβίζουν, τους κρατούν, τους κλέβουν τα υπάρχοντά τους, καμιά φορά τους απολύουν εν τέλει, αλλά πολύ συχνά τους κρατούν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα, η κινέζικη θέση είναι ότι αυτά είναι ψέματα, ότι δεν υπάρχουν. Το πρόβλημα στην Κίνα είναι για τις αρχές ότι υπάρχει το διαδίκτυο, το οποίο επιτρέπει στον κόσμο να αλληλοενημερώνεται. Και υπάρχουν και οι λιγόμενοι bloggers οι οποίοι λένε αυτά τα πράγματα που ισχυρίζεται η ηγεσία είναι γελία. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αυτές οι μαύρες φυλακές. Πρόσφατα ένα κινέζικο παραδοσιακό όργανο, το Outlook του κόμματος. Είπε ότι οι μαύρες φυλακές είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και βάλανε και ένα νούμερο. Ήταν αυστηρότερη από τη δική μας την έκθεση. Υπάρχουν λέει 10.000 10.000 άνθρωποι οι οποίοι πάνε και βρίσκουν τους παραπονούμενους, τους αρπάζουν από τους δρόμους και τους χώνουν στις μαύρες φυλακές. Ήδη οι κινέζικε αρχέ είπαν 10.000. Εμεί δεν είχαμε μπορέσει να βάλουμε νούμερο. Λοιπόν, το, πρόβλημα, το κοινωνικό πρόβλημα είναι τεράστιο. Μία μείζον σύσταση. Εμεί κάναμε μία συνέντευξη τύπου στο Χονγκ Κονγκ, πήγαμε και ε, είχαμε και από το BBC ανταπόκριση και όλου του διεθνεί δημοσιογράφου. Η πίεση, η δημόσια πίεση αποδίδει στην Κίνα και η πίεση με τη δική μας έκθεση και επειδή τέθηκε το θέμα και σε υψηλότερο επίπεδο ως νέο, η, η νέα σας, η κυρία Άστον, η νέα σας είπατε εκπρόσωπος είπε ότι θα το θέσει το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο το δυνατόν συντομότερο να έρθει σε επαφή με τη νέα ύπατη εκπρόσωπο, να είναι σαφέ ότι δεν υπάρχουν ψευδεστήσεις για το τι μπορεί να κάνει κανεί με την Κίνα. Ούτε με διαλόγου, ούτε με σεμινάρια, ούτε με διασκέψεις μπορεί να γίνει πρόοδος. Και σε ό,τι αφορά την θανατική καταδίκη, η μόνη ελπίδα που μπορεί να αποδώσει είναι επειδή τίθεται ξανά και ξανά το θέμα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και με διαρκή πίεση. Μόνο εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμείνει στις αρχές και δημοσίως, οι Κινέζοι ίδιοι μας το λένε, δεν έχει κανένα νόημα να γίνουν τα πράγματα αυτά και κλεισμένων των θυρών. Μόνο δημοσία. Τότε μπορεί να είναι ε, αποτελεσματικό το μήνυμα. Πρέπει να είναι σαφές, ξεκάθαρο και δημόσιο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Άνταμς για τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε ορισμένα θέματα, να υποβάλουμε ορισμένα θέματα στην Βαρόνη Άστον η οποία θα προσέλθει στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η σιωπηλή διπλωματία ως αντιτιθέμενη στην ε, δημόσια πίεση είναι και κάτι το οποίο θα πρέπει να το θέσουμε. Α, ναι, ναι, όχι, συγγνώμη. Η κυρία Άστον θα έρθει αύριο στην Επιτροπή Εξωτερικών. Όχι, όχι στην Υποεπιτροπή μας, αλλά στην Επιτροπή Εξωτερικών. Έχω ένα κατάλογο αγορητών τώρα και έχουμε και άλλους προσκεκριμένους μετά που θα λάβουν το λόγο, πριν από τις 11 πάντοτε. Ο αντιπρόεδρος Σέμκε, ο κύριος Μακμίλαν Εσκότ και άλλα πρόσωπα που είναι παρόντα εδώ. Ο κύριος Ντόμσκι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω όλους του ομιλητές. Ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικέ οι παρατηρήσεις που ακούσαμε. Πάνω απ' όλα όμω, αυτό που με εντυπωσίασε ήταν η ομιλία του κυρίου Βέγγιαν. Ήταν πολύ βαθιά η ανάλυση της κατάστασης των ανθρώπινα δικαιώματα στην οποία προέβη. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες που θα ήθελα να σημειώσω ως προς τις παρατηρήσεις του είναι οι ομοιότητες ε, στις συνθήκες που αντιμετώπισαν οι πρόσπιστες των δικαιωμάτων ε, στην, ε, στο Σοβιετικό μπλοκ πριν από, μερικά, από δύο δεκαετίες ακόμη και τα προβλήματα που βλέπουν και οι Κινέζοι πρόσπιστες των δικαιωμάτων. Και πάντοτε επισήμεναν οι αγοριστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ότι δεν πρέπει να παρασυρθούν οι υπόλοιπες χώρες σε μια υποβάθμιση τη σημασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ούτε να τα παραγνωρίσουν, ε, διότι δεν είναι μια διαφορετική θεώρηση το πρόβλημα. Πρόκειται για ζητήματα τεράστιας σημασίας και κρίσιμα ε, ζητήματα των οικουμενικών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Θα ήθελα λοιπόν ιδιαίτερα να υπογραμμίσω κάποια θέματα, κάποιες ιδέες ιδιαίτερης ευφία του γεγονός ότι δίνει ελεύθερη ε, πρόσβαση, ελευκό επιταγή ε, ο δυτικός κόσμος στην Κίνα με όρους είτε εμπορικούς είτε ασφάλειας. Και επίσης παρά την εξέλιξη της κοινωνίας και ιδιαίτερα την ανάδειξη μιας μέσης τάξης στην Κίνα, τα ανθρώπινα δικαιώματα παραμένουν σε πολύ κακή κατάσταση και εξάγονται σε όρους Λατινικής Αμερικής και Αφρικής ε, σε όλο τον κόσμο. Και εδώ θα σημειώσω εγώ ότι η ιδέα της ε, ελεύθερης οικονομίας της αγοράς, χωρίς όμως τη φιλελεύθερη κοινωνία και τη φιλελεύθερη πολιτική, δεν μπορούν να είναι άλλο παρά ένα εξάμβλωμα και ας μην επιτρέψουμε ούτε στη Λατινική Αμερική, ούτε στην Αφρική, ούτε σε καμιά άλλη χώρα να επαναλάβει το πρότυπο αυτό το οποίο ακολούθησε και επέβαλε η Σοβιετική Ένωση πριν από δύο δεκαετίες. Πρέπει λοιπόν με πολύ μεγάλη προσοχή να, ακολου... ακούμε τους ε, έμπειρους και εμπειριστατωμένους αναλυτές όπως ο κ. Γουενγκιάν. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κύριε Λόχπιλτερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ όλου εδώ παρισταμένου. Έχω μια ερώτηση, η οποία ίσω ξεφεύγει λίγο από τα όσα είπε ο κύριος Βέγγιαν, η οποία μάλλον απορρέει από τα όσα είπε ο κύριο Βέγγιαν, ε, την εμπειρία του και τι ε, ε, παρατηρήσεις που μας διατύπωσε για ένα σεμινάριο του 2008 προς τη συμμετοχή και τη δράση των αγωνιστών για τα ανθρωπινά δικαιώματα. Σε ποιο βαθμό λοιπόν ανταποκρίθηκε στις συστάσεις μας η Επιτροπή από το Ινστιτούτο Πόλτσμαν επίσης ε, θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία που το ε, εκπροσωπεί εάν ε, με ιδιαίτερη εάν μελετούνται οι έρευνες με την ίδια σοβαρότητα από κάθε πλευρά, γιατί θα ήθελα να σημειώσω εδώ ότι τα σεμινάρια ή συστήσεις που κάνουμε εδώ δεν, είναι, δεν πρέπει να είναι μια ευκαιρία να διαφωνήσουμε, αλλά να οξύνουμε το βλέμμα μας ε, ε, ως προς τα θέματα των ανθρωπινών δικαιωμάτων στην Κίνα και αυτό είναι μια σύσταση περισσότερο παρά επίκριση για δε το Ιρλανδικό Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, θα ήθελα να, να παρατηρήσω ότι υπάρχουν, όπως είπατε, κάποιες βελτιώσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τα εξής. Ε, αναφέρατε νωρίτερα ότι υπάρχει η μία τάση, ξεκινάει μια νέα διαδικασία στην Κίντα ως προς την, ε, κατάρ, κατάργηση της θανατικής ποινής ε, για εγκλήματα που δεν είναι βία ή να περιοριστεί εν πάση περιπτώσει η πολύ θανατικής ποινής. εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα τέτοιο, θα ήθελα να μου δώσετε περισσότερα στοιχεία. Και δεύτερον για τα δικαιώματα των πολιτών. Υπάρχουν κινήματα από ό,τι ισχυρίζεται η Κίνα, αλλά είναι σε θέση η κυβέρνηση, η διοίκηση να παρεμβαίνει σε, περι... σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εάν βλέπετε κάποια εξέλιξη ως προς την επιβολή αυτών των διοικητικών κυρώσεων, δηλαδή του διοικητικού περιορισμού της ελευθερίας, ε, εις βάρος τέτοιων αγωνιστών των δικαιωμάτων. Πολλές φορές μάλιστα ε, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αναπτύσσουν δραστηριότητα ως πολίτες, όχι μόνο σε άγνωστες ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά μέσα στην κοινωνία τους όσοι δραστηριοποιούνται, αντιμετωπίζουν ε, μεγάλη μεγάλες δυσκολίες και μας λένε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται από τη δική μας την πλευρά να συζητήσουμε τα προβλήματα αυτά, τους βοηθούν γιατί βρίσκουν περισσότερη ανταπόκριση μέσα στις κοινωνίες Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ανδρικίενε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστώ και εγώ όλους τους ομιλητές που έλαβαν το λόγο σήμερα. Ήταν άκρος ενδιαφέρουσες οι εισηγήσεις σας, πολύ ενημερωτικές. προφανώ εδώ εμεί γνωρίζουμε αρκετά καλά τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα γιατί τα παρακολουθούμε εδώ και καιρό. Υπάρχουν διάφορε εκδηλώσει. όπως μια ακρόαση που είχαμε και πρόσφατα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα. Ξέρετε ότι τα θέματα αυτά το Κοινοβούλιο τα παρακολουθεί εδώ και καιρό. Είναι ένα όργανο θεσμικό το οποίο εδώ και πολύ καιρό έχει υψώσει τη φωνή του και μιλάει δυνατά για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα δεν μπορεί κανείς να υποχρεώσει το κοινοβούλιο μας να αγνοήσει ή να, αλλά να αγνοήσει τα προβλήματα ή να αλλάξει στάση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα. Δεύτερον, ως προς το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα σεμινάρια. Είχα την ευκαιρία πριν από ένα χρόνο περίπου, επισκεπτόμενη την Κίνα σε, με μια αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου, να, συζητάς να συζητήσω τα θέματα αυτά. Ε, υπήρχε εκείνη την εποχή ένα σεμινάριο στην Κίνα και την τελευταία ημέρα του σεμιναρίου επισκέφθηκε η αντιπροσωπεία μας και ενημερώθηκε ότι ένας Κινέζος υπήκος ο οποίος είχε ενυμφευθεί μια Αυστριακή ε, είχε κατηγορηθεί για κατασκοπία και καταδικαστεί σε θάνατο. Ήταν η τελευταία ημέρα αυτή τη επαφή, αυτού του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου ήρθε η είδηση για την ε, καταδίκη σε θάνατο. Πέρυσι επίσης είχαμε το θέμα των Ουιγούρων ε, και άλλων που καταδικάζονταν ομάδικα σε, ε, στην θανατική ποινή. την εποχή ακριβώ που αναπτυσσόταν ο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτέ λοιπόν οι βίες καταστολέ ή η επιβολή θανατική ποινή ακριβώ την εποχή κατά την οποία αναπτύσσεται ο ε, διάλογος διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για μένα δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά προκλήσει από πλευρά του καθεστώτο τη Κίνα. Κάθε φορά δηλαδή που θέλουμε να συνομιλήσουμε με κάποιον αγωνιστή για τα δικαιώματα του ανθρώπου, τον απειλεί ε, η θανατική ποινή. Μόνο ένας στόχο μπορεί να υπάρχει, ε, να εξυπηρετείται από το γεγονός αυτό. Να ε, μην συζητηθούν τα πιο ευαίσθητα ζητήματα ή να ξεχάσουμε ποιος είναι ο στόχος μας. Να χαθεί δηλαδή η ουσία του διαλόγου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αναδιατυπώσουμε την στρατηγική μας για την Κίνα και θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις συστάσεις των περισσότερων των ομιλητών των εδώ Σε Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενο ομιλητή. Θα πω πρώτα ότι υποστηρίζω πολύ τα όσα μας είπατε σήμερα και σας ευχαριστώ πολύ και την τεκμηρίωση που μας έχετε προσφέρει. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, και που είπε κάποιος προηγουμένως, η κυρία Αντρικένε μάλιστα, ότι χρειάζεται να επανεξετάσουμε τους στόχους μας και τη στρατηγική μας. και το τι γίνεται ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κίνα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι το χειρότερο ενδεχόμενο που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε θα είναι να συζητούμε κάπου κάπου, να κάνουμε ιδιαίτερα εξόχως ενδιαφέρουσες συζητήσεις, αλλά οι συζητήσεις αυτές να αποδίδουν πολύ μέτρια αποτελέσματα. Νομίζω ότι αυτό που καλούμαστε να κάνουμε εδώ είναι να είναι πραγματικά χειροπιαστά αποτελέσματα. Γι' αυτό το λόγο καταβάλουμε την προσπάθεια αυτή. Η δουλειά μας είναι να βελτιώσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα. Όχι απλώς να καθόμαστε και να συνομιλούμε. Πρώτο πρόβλημα λοιπόν Πρώτο ερώτημα. Η Κίνα είναι ανοιχτή να συζητήσει το ενδεχόμενο ανάληψη δράση που να είναι σύμφωνε με αυτά που επιθυμούμε. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η Κίνα γνωρίζει καλά την δύναμή τη. Γνωρίζει καλά ότι είναι παραπάνω από το διπλάσιο της Ευρώπης Η Κίνα γνωρίζει επίσης καλά ότι υπάρχουν χώρες που μιλούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες τηρούν σιγή και προτιμούν τις business. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε πίεση στην Κίνα. η Κίνα δεν είναι πλέον απομονωμένη. Η Κίνα ε, έχει, συνεργάζεται και έχει να αντιμετωπίσει ένα πλήθος άλλων χωρών. Άρα πρέπει να λάβει υπόψη της το τι γίνεται και το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο και τι ζητούν οι άλλες χώρες. Εν προκειμένου, νομίζω ότι μπορούμε να διατυπώσουμε τρεις συστάσεις. Πρώτη, εμείς εδώ στην Ευρωβουλή έχουμε φτάσει σε ένα χρονικό σημείο το οποίο ε, είναι σημαντικό διότι θα έχουμε σύντομα νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προβλέπεται ακρόαση με την ε, νέα ύπατη εκπρόσωπο εξωτερικής πολιτικής. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να ζητήσουμε από την ε, νέα ύπατη εκπρόσωπο είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα να περιληφθούν σε όλους τους τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να γνωρίζουμε σαφώς ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ευκαιριακά. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός τομέας και θα πρέπει να μπουν στον πυρήνα και στην καρδιά όλων των δράσεών μας. Είναι η πρώτη θητεία μου ως Ευρωβουλευτής. Εγώ έχω περάσει από το Πολωνικό Κοινοβούλιο πρώτα. Αλλά θέτω το εξή ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναπτυχθεί, θα αναπτύξει και τα γραφεία εκπροσώπησής της σε, όλη, σε όλο τον κόσμο. Ασκώντας μια διπλωματική δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο. Διερωτώ πόσο ισχυρή θα πρέπει να είναι η εντό εισαγωγικών πρεσβεία μας στην Κίνα. Ίσως πρέπει στην πρεσβεία μας στην Κίνα να έχουμε να περιλάβουμε μια μονάδα η οποία θα ασχολείται ειδικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα. υπενθυμίζω για ποια πράγματα μιλούμε. Μιλούμε για την θανατική ποινή στην Κίνα. Και η προσέγγιση μας είναι πολύ διαφορετική. Είπε κάποιο σήμερα ότι όλο και περισσότερες θανατικές ποινές εκτελούνται. Ένας άλλος ομιλητής όμως είπε ότι υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις. Έχετε υπόψη σας όμως τους κώδικες προβλέπει η θανατική ποινή, απειλεί τη θανατική ποινή για 68 αδικήματα. Ακόμα δηλαδή και παράνομες επιχειρηματικές δραστηριότητες μπορεί να τιμωρηθούν με την θανατική ποινή. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κ. Σάμπας, ότι διατρέχουμε σοβαρό κίνδυνο προσπαθώντας να επιτύχουμε ταυτόχρονα πολλούς στόχους. Αυτό που χρειάζεται είναι να ρίξουμε ιδιαίτερο βάρος σε βασικά θέματα, σε θεμελιώδη θέματα όπως αυτά που άπτονται τη ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε Ζέμκε. Τέσσερις συνάδελφοί μου βρίσκονται και γραμμένοι στον κατάλογο των αγοριτών. Αν θέλουμε να ακούσουμε απαντήσεις από τους ε, προσκεκλημένους μας, θα σας παρακαλέσω όλες και όλους να μιλήσετε σύντομα, το πολύ ένα λεπτό ο καθένας ή η καθεμία, για να έχουμε χρόνο για απαντήσεις. Μακμίλαν Σκοτ, Πρέβρος και θα ακολουθήσουν άλλοι δύο. Σεις, κύριε Μακμίλαν Σκοτ. Ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Ξέρετε, Πρόεδρε, ότι μου ανέθεσε ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου υπό την ιδιότητά μου ω ε, αντιπρόεδρο να παρακολουθώ τα θέματα των σχέσεων όλων των θεσμικών οργάνων εν ώψη της, του ελέγχου των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Εγώ επισκέφθηκα την του 2006 και όλοι οι ε, αντικαθιστωτικοί, όλοι εκείνοι που αγωνίζονταν για την μεταρρύθμιση του καθεστώτος βρίσκονταν στη φιλική όσο πιο ζήτησα να δω ε, πολλά ονόματα σας απαριθμό που δεν μπόρεσα να συναντήσω γιατί βρίσκονταν στη φυλακή. Συνεχίζονται για πολλούς από αυτούς και η φυλάκιση και οι βασανισμοί αλλά γενικά συνεχίζεται και η κακή κατάσταση στην Κίνα και παρά ή πέραν του βραβείου Ζαχάροφ, που βεβαίως έχει μεγάλη απήχηση, πέρυσι απενεμήθη στον Γουτζά, βρισκόταν ε, φυλακισμένος και ταυτόχρονα με την απονομή αναφέραμε και πολλούς άλλους ε, ε, φυλακισμένους αντικαθεστατικούς. Πέραν λοιπόν αυτής της διαδικασίας του βραβείου Ζαχάροφ, μπορούμε ε, να έχουμε τη διαδικασία Salzgitter και έχω εδώ το βιβλίο, το οποίο, μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει από την ε, Ανατολική Γερμανία και που επιτρέπει σε έναν κρατούμενο, έναν φυλακισμένο, έναν βασανιζόμενο να πει στον δεσμοφύλακά του, στο βασανιστή του, ε, ότι κοίταξε, εγώ σε έχω καταδώσει και το όνομά σου θα το λάβει η οργάνωση Salzgitter. Ιδιαίτερα από την Κίνα, αλλά και από πολλέ άλλε χώρε, που υπάρχουν ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μπορούμε, πιστεύω, να συλλέξουμε τον τρόπο αυτό στοιχεία. Πρόκειται για μια οργάνωση την οποία υποστηρίζει και μπορεί να χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία στρέφεται ακριβώς εναντίον τυραννικών ε, καθεστώτων όπως αυτού της ε, Κίνας ε, και μπορεί να προσφέρει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση και στη βελτίωση των συνθήκων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τρόπο που δεν μπορεί να εξασφαλίσει, παραδείγματι, η Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών λόγω των περιορισμών που επιβάλλει το Συμβούλιο Ασφαλείας με το σύστημα ψηφοφορία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω συγκεκριμένες ερωτήσεις προς την Επιτροπή. Σχετικά με τις διακρίσεις κατά των θρησκευτικών μειονοτήτων στην Κίνα. Τι γίνεται με τους γιουγούρους. όπου τα δικαιώματά τους έχουν περιοριστεί και δεν γίνεται τίποτα για να βελτιωθεί η κατάσταση. Θα ήθελα να ξέρω τι έκανε η Κομισιόν. Έγιναν δηλώσεις του Συμβουλίου για τις, κατά των εκτελέσεων, αλλά οι εκτελέσεις παρόλα αυτά γίνανε. η Κίνα μου απάντησε ότι η Κίνα μάλλον απάντησε ότι εκκρεμούν ακόμα δίκες και θα ακολουθήσουν και άλλες εκτελέσεις. Η Κομισιόν λοιπόν τι σκοπεύει να κάνει. Πώς προτίθεται να μεσολαβήσει. Θα είχα και άλλες ερωτήσεις ε, για τους εμπειρογνώμονες, αλλά ο χρόνος μου είναι περιορισμένος και σταματάω με αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κούκαρα έχει το λόγο, χωρίς μικρόφωνο. I really appreciate all the Ιδιαίτερα θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για όλες τις πληροφορίες που λάβαμε σήμερα εδώ με τη συζήτηση. είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ωστόσο, όπως είπε ο κύριος Ζένκα, έτσι και εγώ βλέπω ότι η ανάλυση, οι πληροφορίες, οι συζητήσεις, ε, ο διάλογος, λόγο έχουν, σκοπό έχουν να εξασφαλίσουμε την πιο αποτελεσματική στρατηγική για τον τρόπο αντιμετώπισης ε, των επισήμων φορέων των αρχών της ε, Κίνας έτσι ώστε να τις πείσουμε να βελτιώσουν θήκε προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και σεβασμού των ανθρώπων. Διαφορετικά περιοριζόμαστε μόνο σε μια ακαδημαϊκή συζήτηση και γι' αυτό ιδιαίτερα ευχαριστώ την κυρία Κίνσελμπαχ για τις ε, παρατηρήσεις σας και ιδιαίτερα ε, την εύστοχη προσέγγιση του κυρίου Άνταμς. Μπορεί να είναι αφελής για τους λοιπούς η παρατήρησή μου, αλλά θα τη διατυπώσω παρόλα αυτά. Είπε λοιπόν ο κύριος Άνταμς ότι η ήπια, η, η ήσυχη διπλωματία ίσως είναι πιο αποτελεσματική από την ε, ανοιχτή και δημόσια πίεση. Θα αποκλείεται κύριε Άνταμς το συνδυασμό των δύο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ο ε, κύριος Χάουιτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ για την κυρία Κίνσιλμπαχ. Εδώ είμαι, εδώ Δεν αντιλαμβάνομαι πώς είναι δυνατόν να ισχυρίσετε κανείς ότι υπάρχει χώρα από την οποία... Εδώ στα δεξιά σας είμαι, καλημέρα σας. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να λέτε ότι μπορεί κάποια χώρα Εντάξει, οικονομικές κυρώσεις μπορώ να φανταστώ, άλλες συμβολικές κυρώσεις κλπ. Αλλά να αποχωρήσουμε από το διάλογο για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Πώς είναι δυνατόν. Άκουσα τις επικρίσεις ε, που διατυπώθηκαν σε βάρος αυτής της ε, πρότασης. Δεν καταλαβαίνω τι χρησιμότητα θα έχει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό παρακαλώ να μου εξηγήσετε περισσότερο, γιατί αμφισβητώ πολύ την κρίση σας αυτό. Για τον κύριο Σαμπάς, καθηγητή Σαμπάς γιατί υπήρξε αυτή η κινητικότητα προ θερατική ποινή. Είπατε ότι υπήρξε κάποια εξέλιξη. Ναι, αλλά πρέπει να δούμε πού ακριβώ είναι το κουμπί που θα ε, πιέσει την κινέζικη κυβέρνηση να προχωρήσει ακόμη περισσότερο στο διάλογο και σε ουσιαστικέ μεταρρυθμίσει. Με ποιο τρόπο μπορούμε να του επηρεάσουμε. Αυτό θέλουμε εσεί να μα προσφέρετε. Πού ακριβώ βρίσκεται η... το σημείο πίεση. Δεν έχω πολύ χρόνο όμω. Δεν θα ήθελα καλά να πω, αλλά περιορίστω σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χάουετ. Θα πρότεινα το εξή για να οργανωθούμε, για να οργανώσουμε το χρόνο μας. Ο κύριος Μέτεν, επίσης προσκεκλημένος μας ε, από την ε, εκστρατεία για την απελευθέρωση του Θιβέτ, θα μπορούσε να λάβει δύο λεπτά για να μας μιλήσει ε, και στη συνέχεια να επανέλθουμε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή που θα μας ε, δώσουν τις δικές τους προτάσεις και παρατηρήσεις. Vincent Metten, παρακαλώ, από την Εκστρατεία για την Απελευθέρωση του Θιβέτ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Από το Μάρτιο του 2008, 235 ειρηνικές διαδηλώσεις κατά την πλειοψηφία έγιναν στο Θιβέτ. Και η καταστολή επικρατεί σε όλο το Θιβέτ. Σήμερα λοιπόν στο Θιβέτ υπάρχει ένα πάρα πολύ άσχημο κλίμα, ένα τεράστιο άγχος στον πληθυσμό και η Κίνα παίζει το επικίνδυνο χαρτί του εθνικισμού. 735 κρατούμενοι από το Μάρτιο του 2008 και 1200 νοούμενοι. Plusieurs personnes ont reçu de longues peines de prison et beaucoup de personnes Έχουν γίνει καταγγελίες για βασανιστήρια. Αλλά δεν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες, διότι οι αλλοδαποί δεν μπορούν να πλησιάσουν στην περιοχή. Οτιδήποτε εκφράζει την θηβετιανή ταυτότητα, την πολιτιστική ταυτότητα, την κουλτούρα του Θιβέτ καταστέλλεται. Όμως, παρόλα αυτά, διανοούμενοι, συγγραφείς, ε, bloggers συνεχίζουν να αντιστέκονται. Ορισμένοι από αυτούς έχουν εξαφανιστεί, έχουν φυλακιστεί. Πέντε φιβετιανοί έχουν καταδικαστεί σε θάνατο. Από αυτούς τους πέντε, δύο έλαβαν, ε, τρεις έλαβαν αναστολή και δύο εκτελέστηκαν. Η οργάνωσή μας ασχολείται ιδιαίτερα με τα βασικά και, και την αυθαιρεσία των της κινέζικης δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής δικηγόρου, ο χρόνος της δίκης είναι, της προφυλάκησης συγγνώμη, είναι περίεργα ρυθμισμένος, δεν υπάρχει πληροφόρηση προς τις οικογένειες, δεν ξέρουμε πώς εξελίσσεται η δίκη και οι ξένοι διπλωμάτες επίσης δεν ενημερώνονται. Εμείς θα θέλαμε να έχουμε μία, την εγκρισή μία ενιαίας πολιτικής για το Θιβέτ για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια. Θα έπρεπε να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών και της Κίνας για αυτά τα θέματα. Και αν κατά τη διάρκεια του διαλόγου συνεχίζεται η κινέζικη αδιαλαξία, αυτή η αδιαλαξία θα πρέπει να αναφέρεται και στο τελικό πρακτικό των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή στη διάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας θα πρέπει να φαίνεται σαφώς η διαπλοκή με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μέτινα. Άλλωστε έχουμε και τη γραπτή σας ε, δήλωση. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, συζητήσαμε το θέμα του Θιβέτ ε, και το, με το ψήφισμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο και πάλι στον προσευτή κύριο Νόρτλαντερ για σύντομες παρατηρήσεις για να επανέλθουμε μετά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες ε, οι παρατηρήσεις και οι απόψεις τους. Θα ήθελα να σημειώσω ότι η Προεδρία αλλά και όλοι μας ανησυχούν ιδιαίτερως για, τις, ε, για την τύχη του κυρίου Γκυλγκόρ και του, του κυρίου Γκάου Σέγγ που αναφέρθηκαν νωρίτερα. τον στον ε, διάλογο αυτό σημειώνουμε ανησυχία για την τύχη του δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση, αλλά πιστεύουμε ότι η δική του η περίπτωση έχει ύψιστη σημασία. Και θα ήθελα, Πρόεδρε, να πω μερικά λόγια για τον διάλογο και τη χρησιμότητά του. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο, ίσως και αδύνατο να προσμετρηθεί η σημασία ή ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει αυτός ο διάλογος. Ας φανταστούμε όσο θα γινόταν εάν δεν υπήρχε διάλογος. Εάν δεν υφίστατο καν. Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω τα λόγια κάποιου εκ των οικοδεσποτών μας από μια αρσιατική χώρα στον, ε, σε μια εκδήλωση που είχαμε. Μετά την συζήτηση και στο δείπνο που είχαμε με τους Ασιάτες οικοδεσπότες μου είπε λοιπόν ο κύριος αυτός δεν άκουσα ποτέ κανέναν ε, να προβάλλει επιχειρήματα, να μιλάει όπως εσείς και να προβάλλει τα δικαιώματα κατά τον τρόπο που τα προβάλλετε εσείς. Δεν θα ήταν λοιπόν σωστό πιστεύω να υποβαθμίζουμε τη σημασία της επικοινωνίας με τους άλλους, του να μιλούμε με τους άλλους ανθρώπους, γιατί οι ανθρώπινα δικαιώματα είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη προστασία τους από την πυθό που μπορούμε να ασκήσουμε, από την ανθρώπινη επαφή που μπορούμε να αναπτύξουμε. Χρειάζεται φυσικά μεταρρύθμιση σημαντική και πολλά ακόμη έχουμε να κάνουμε εμείς για να συμπεριλάβουμε τις έννοιες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με βάση αυτά να ε, ε, προβαίνουμε στην σύναψη και εκτέλεση συμφωνιών σε κάθε τομέα πολιτικής. Το ίδιο πιστεύω το αναφέρουμε και στο ανακοινωθέν ε, από τον διάλογο Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας ότι ε, πρέπει να γραφούν και μέσα στον πολιτικό διάλογο. Δεν μπορούμε όμως να περιοριστούμε μόνο στον πολιτικό διάλογο διότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ένα τομέα ανάπτυξης επιχειρημάτων που δεν μπορούν να αποτελούν ένα τομέα τόσο ευρύ που δεν μπορούν να καλύψουν με τα επιχειρήματά τους ή μέσα στο διάλογο τους οι πολιτικές μας αρχές. Και γι' αυτό ε, απαραίτητο είναι να διαφυλαχθούν όλα τα μέσα που έχουμε στη θέση μα. Όχι μόνο ο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όχι μόνο ο πολιτικό διάλογο, αλλά όπω υπόθηκε νωρίτερα, οι αντιπροσωπείε μας, οι διπλωματικές αποστολές στο Πεκίνο. Όλες οι εκδηλώσεις οι συναντήσεις ε, που έχουμε και θα ήθελα να πω ότι κατά τη δική μας την Προεδρία μόνο αυτό το φθινόπωρο είχαμε επτά διαφορετικές ε, ευκαιρίες ε, με αντιπροσωπείες, ε, συζητήσεις, διαβήματα, διάλογο, να μιλήσουμε με τις κινέζικες αρχές στο Πεκίνο. Ήταν πολύτιμες ευκαιρίες, ευκαιρίες που αξιοποίησαμε στο βαθμό που μπορούσαμε και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο στον ε, διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και έτσι αναγνωρίζω ότι όντω είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να βελτιωθεί έτσι περαιτέρω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή παρακαλώ. One comment to complement what Ambassador said. I mean, there is no doubt. Μια μικρή συμπλήρωση στα όσα είπε ο πρέσβης. Ασφαλώς δεν μπορεί κανείς να ακολουθήσει μία μοναδική και ενιαία οδό για ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που έχουμε ε, απέναντι στην Κίνα. Έχουμε και σημαντικά προβλήματα σε άλλους τομείς. Εμπόριο, ε, αλλαγή κλίματος κλπ. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι ηγέτες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να βρουν τη σωστή ισορροπία ανάμεσα σε όλα αυτά τα θέματα. Βεβαίω, τα ανθρώπινα δικαιώματα παραμένουν μια σημαντική παράμετρο, αλλά να εκφράσουμε τι ανησυχίε μα στου Κινέζου. Και όπως είπε ο κύριος Πρέσβης, χρησιμοποιούμε ένα συνδυασμό δημόσιας πίεσης και α, σιωπηρής διπλωματίας. Που ορισμένοι θα πούν βέβαια ότι δεν είναι ε, αποτελεσματική. Όμως νομίζουμε ότι τα μηνύματά μας περνούν και γίνονται κατανοητά. Για τον ίδιο το διάλογο τώρα, η αξιολόγηση συνεχίζεται, οι συζητήσεις συνεχίζονται δεν είναι ανάγκη λοιπόν τώρα να προσπαθήσουμε να προκαταλάβουμε τα αποτελέσματα των συζητήσεων αυτών. Ωστόσο, συστηματικά έχουμε παρακολουθήσει όλα τα θέματα. Δεν υπάρχει εμφιβολία ότι έχουν σημειωθεί βελτιώσεις όπως είπε και ο καθηγητής Σάμπας. Υπάρχουν νέοι νόμοι καλοί. Ασφαλώ η υλοποίησή του στο τοπικό επίπεδο έχει κενά. Δημοσιεύσαμε και το νέο σχέδιο δράσεως για τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι και σημαντικό benchmark για να δούμε στα ε, τέλη της διετίας που έχουμε δώσει τι θα έχουν επιτύχει, αλλά το πιο σημαντικό και ας μην το λησμονούμε είναι ότι ο διάλογος ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας επιτρέπει να θέτουμε με ε, ιδιαίτερη έμφαση όλα τα θέματα. Και νομίζω ότι έχουμε κάνει αυτό συστηματικά και ταυτόχρονα όπως κάναμε για τις άδειες ασκήσεις επαγγέλματος των ε, συνηγόρων. Αυτή τη στιγμή το πράττουμε και σύμφωνα με όλες τις στατιστικές μας είναι καλύτερη η μεταχείριση που τους επιφυλάσσεται μετά. Άρα είναι ένα σημαντικό, μια σημαντική παράμετρος που δεν πρέπει να τη λησμονούμε. Και δύο πιο συγκεκριμένα ερωτήματα που τέθηκαν. Για την δίκη για τις δίκες και για τις, ε, ε, για τις δίκες, δίκες ε, των ουγούρων, ναι, των ουγούρων. ζητήσαμε να είναι δίκες, οι δίκες βεβαίως υπήρξε κάποια ανταπόκριση. Τώρα γίνεται, από την, γίνεται το σεμινάριο διοργάνω το σεμινάριο από το Πανεπιστήμιο του Γκόρουι και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και ευγνώμονε για την βοήθεια που λαμβάνουμε από το όργανο αυτό. Σα ευχαριστώ, ε, Επιτροπή. Κύριε Γουενκιάνγκ, εσεί τι λέτε για αυτή τη συζήτηση. Θα μεταφράσει η συνάδελφός μου, θα μιλήσω κινέζικα. Θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια, απαντώντα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχόλιο που έκανε για το σχέδιο δράσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δημοσίευσε η κινέζικη κυβέρνηση. Στην Κίνα χρησιμοποιούμε ένα γνωμικό που λέει τα έργα είναι καλύτερα από τα λόγια. Όντως, το σχέδιο δράσεως ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δημοσίευσε η κινέζικη κυβέρνηση δημοσιεύτηκε από την ε, κινέζικη κυβέρνηση το σχέδιο δράσεως εκδόθηκε από την κινέζικη κυβέρνηση στο χρονικό περίπου διάστημα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008 με στόχο να βελτιωθεί η εικόνα προς τα έξω της Κίνας. Μετά από την έκδοση του σχέδιου δράσεως, μετά από τη δημοσίευσή του, η κατάσταση των οποίων δικαιωμάτων στην πραγματικότητα επιδεινώθηκε στην Κίνα. Και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Kiitos tästä lyhyestä ja selkeästä kommentista, herra Venkian. Sitten... Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ξεκάθαρη δήλωση. Ο κύριος Κιλγκόρ. Μικρόφωνο παρακαλώ, μικρόφωνο. Το 2004 υπήρξαν 3.400 εκτελέσεις και αυτές μειώθηκαν κατά ορισμένες εκατοντάδες μετά τα επόμενα χρόνια. Αλλά πρόσεξα ότι ο πρόσωπος της Κομισιόν δεν μίλησε καθόλου για το Falun Gong. Δεν εμφανίζονται ε, τα νούμερα των οπαδών του Falun Gong που θανατώνονται και τα όργανά τους επαναχρησιμοποιούνται. Δεν είπε τίποτα. Ο καθηγητής Μπέρντεν πρότεινε ο ίδιος ε, πρώην διπλωμάτης να σταματήσουμε τον διάλογο. Και θέλω επίσης να αποτίσω ιδιαίτερο φόρο τιμής για τον στον Σκότ, ο οποίος είναι ακούραστος εργάτης στην υπόθεση του ε, Φαλουνγκόγκ. Και εσείς κύριε καθηγητά Σάμπας, δεν, μπορεί, δεν μπορούμε να στερούμε θα σπονδυρική στήλη για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κιλγκόρ. όσοι παρακολουθούν τα θέματα της Κίνας γνωρίζουν ότι υπάρχουν θέματα ταμπού όπως η δυτική χώρα, το Θιβέτ και η Φαλούν Κόγκ. Δεν επιτρέπεται δηλαδή να συζητηθούν με τις αρχές της Κίνας. Εσείς επίσης κύριε Κισελκάρτ ε, ακούσατε πολλές παρατηρήσεις ε, που υποθύνονταν σε εσάς. Θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ όλους όσοι διατύπωσαν παρατηρήσεις ε, και που μου επιτρέπουν έτσι να διευκρινίσω κάποια σημεία. Ε, ρεαλιστικά, διάλογο πρέπει να διατηρήσουμε, δεν πρέπει να σταματήσουμε ποτέ να μιλάμε. Εγώ δεν είπα ότι πρέπει να σταματήσουμε το διάλογο. Είναι πολύ σημαντικό το να συζητούμε, αλλά πρέπει και ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει ποιο διάλογο φέρνει αποτελέσματα και ποιο δεν φέρνει αποτελέσματα. Εγώ δεν προτείνω να σταματήσει ο διάλογο με την Κίνα. Είπα να σταματήσει τουλάχιστον να περιοριστεί η διεξαγωγή διαλόγου σε ένα περιορισμένο περιθωριοποιημένο πλαίσιο μόνο μεταξύ κάποιων αξιωματούχων. Εδώ έχουμε να κάνουμε ουσιαστικά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το να ε, περιμένει κανεί ότι ένα τέτοιο περιθωριοποιημένο διάλογο μπορεί να προσφέρει αποτελέσματα και αλλαγέ στην Κίνα είναι μη ρεαλιστικό. Πρέπει ο διάλογο να επανέλθει στην κοινή γνώμη. Πρέπει να επανέλθει στο δημόσιο πεδίο. Σας ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ. Και εγώ ενστερνίζομαι με το είπε η Κάθριν Κιντζιλμπαχ. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι διάλογος υπάρχει πάντοτε, όπω και αν τα πράγματα. Ε, πρέπει να δούμε όμως εάν το αποτέλεσμα που φέρνει είναι προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή περιθεωροποίησή του. Ανάλυση δεν έχουμε κάνει για να καταλήξουμε σε ένα από το συμπέρασμα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να, να προσέξουμε την πτυχή αυτή. Διάλογο θα υπάρχει. Διμερή θα είναι, διπλωματικό θα είναι, πολιτικό θα είναι, πολυμερή θα είναι, διασκέψει, συζητήσει μεταξύ επιστημόνων, νομικών, ελευθερία τη άποψη. Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα στην Κίνα διαρκώ. Το θέμα είναι αυτό ο διάλογο. Ο διάλογο με άλλε χώρε προσφέρει αποτέλεσμα. Και για να προχωρήσω ακόμη προ το ζήτημα τη ε, διπλωματίας, της σιωπηλής διπλωματίας. Ναι, βεβαίως, δεν μπορεί να παραμείνει μόνη προσέγγιση, γιατί πρέπει αυτή την ήσυχη ήπια διπλωματία να τη συνοδεύει και μια στεναρή δημόσια τοποθέτηση. Και εδώ αυτό πιστεύω θα πρέπει να προσέξουμε να ε, επαναφέρει τα ανθρώπινα δικαιώματα ως ύψιστη προτεραιότητα στο χώρο συζητήσεων. Γιατί πολλές φορές, ύστερα από μια διάσκεψη, βγαίνει το ανακοινοθέν το οποίο λέει Α, ναι, συστήθηκαν και τα ανθρώπινα δικαιώματα και μετά ανακαλύπτουμε ότι μόνο δύο λεπτά είχαν αφιερωθεί προ το τέλο τη συζήτηση στο θέμα αυτό. Όχι, πρέπει να επανέλθουν στο επίκεντρο των συζητήσεων. Επίση, μιλήσατε για την σχετικότητα τη διαδικασία του διαλόγου. Κάποιο μίλησε από κυριαρχική πλευρά για ένα πρόβλημα σχετικό με, ένα, με την ανέγερση ενό μουσουλμανικού τεμένου στη Σουηδία ω παράδειγμα προβλημάτων ανθρώπινων δικαιωμάτων Σουηδία. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε, γιατί πρέπει να δίνουμε την απάντηση και να επανερχόμαστε με μία σειρά ε, ερωτήσεων που θα μιλούν για τεμένη στην Κίνα. Όχι ελευθερία τη ε, έκφραση ή το δικαίωμα στην αναφορά. Θέλετε να μιλήσουμε για τεμένη. Πολύ καλά. Ανοίγετε το θέμα του τεμένου στην ε, Σουηδία. Θα ανοίξουμε και εμεί το θέμα των τεμενών στην Κίνα. Όπω είπε και ο κύριο Βέγγεν Τζάου. υπάρχει μια πάγια πολιτική, μια ε, επιλογή του καθεστώτος που δεν επιτρέπει την ανέγερση τεμενών ή την προαγωγή του, της θρησκείας, της πιο αδύναμης κοινότητας, της πιο, ε, ε, του πιο περιορισμένου αριθμού ανθρώπων, της κουλτούρας ή της θρησκείας ή του τρόπου σκέψης κάποιου διαφορετικού. Αυτό λοιπόν νομίζω θα πρέπει να προβληθεί και θα ήταν μια ενδιαφέρουσα αλλαγή. Επίση, θα ήθελα να σημειώσω ότι πρέπει να θυμάστε πάντοτε ότι το πρόβλημα για του Κινέζους δεν είναι ούτε το κέντρο τη Ιρλανδίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή ε, ότι μπορεί να ζητάτε κάποιε βελτίωσει εσεί. Εγώ δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει η οτι μπορει να ζητατε καποιε βελτιωσει εγω δεν γιατί το, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στην ευρωπαϊκή πλευρά. Το θέμα είναι αν οι Κινέζοι θα μπορέσουν να επιφέρουν τι αλλαγέ. Αλλά πρέπει αυτό κάθε φορά να το ζητάμε, να το προβάλλουμε. Οι Ιρλανδοί καημένοι στον κόλπο ούτε καν ξέρουν. Την άλλη μέρα έχουν συνεδρίαση, έχουν συνάντηση επιστημονική και δεν ξέρουν αν θα λάβει χώρα καν. Ε, αυτό όλο πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστώ, ο κύριος Σάμπας. Καθηγητής κύριος Σάμπας. Ποτέ δεν με αποθάρρυναν οι δυσχέρειες των ε, θεμάτων Νομίζω ότι είναι υπερβολικό να πει κανεί ότι είναι απόλυτα μονομερές και ότι ε, οι συναντήσεις αυτές δεν έχουν αποδώσει και στον διάλογο και σε άλλες παρόμοιες δραστηριότητες όπως ε, το project για την θανατική καταδίκη ε, από το Βρετανικό Κέντρο Κίνας ή έχουν νόημα και αποδίδουν. Είναι κάπως σαν να προσπαθούμε να δείξουμε και πάλι μιλώ για την πανεπιστημιακή πλευρά, για το νομικό σεμινάριο, σαν να προσπαθούμε να καταδείξουμε Ορισμένοι θα πούν ότι στην πραγματικότητα εμείς ε, συζητούμε και τα πράγματα έξω στον κόσμο γίνονται διαφορετικά. Νομίζω ότι ο κύριος Χάουιτ ρώτησε αν γνωρίζουμε για ποιο λόγο υπήρξε κάποια μείωση των θανατικών καταδικών. Υπήρξε τα τελευταία κυρίως δύο χρόνια μείωση των θανατικών εκτελέσεων. Είναι μεγαλύτερος αριθμός πάντως θανατικών εκτελέσεων και από όλους, όλες όσες γίνονται στον κόσμο. Τα είπαν αυτά και στα Ηνωμένα Έθνη και στο Συμβούλιο της Ευρώπης έχουν κάνει μια, μια προσπάθεια. Το ίδιο όμως και οι, καταδί... και οι καταδίκες των θανατικών καταδικών και ούτω καθεξής. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι, ε, διαφωνεί κανένας, αυτοί δηλαδή που επιχειρηματολογούν υπέρ του διαλόγου, είτε είναι και πανεπιστημιακοί και κάθονται και συζητούν, δεν αμφισβητούν το γεγονός πάντως ότι η δημόσια καταδίκη των πρακτικών αυτών ασφαλώς έχει ένα ρόλο να παίξει υπό ορισμένε συνθήκες και δεν θέλουμε να εξαφανιστεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι ήσυχε ε, συζητήσεις και οι ε, πανεπιστημιακές ανταλλαγές δεν ε, συνεισφέρουν και αυτές. Ο κ. Ντόνσκης έκανε μια ε, αναλογία με ε, πολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη. Είμαι βέβαιος ότι τα τέλη της δεκαετίας του 70 και του 80 θα είχαμε τις ίδιες συζητήσεις, εάν δηλαδή η, η σιωπηλή η διπλωματία και οι συζητήσεις των πανεπιστημιακών που γίνονταν της Συμφωνίας του Ελσίνκη απέδωσαν κάτι. Αυτό που θα το συζητήσουμε ακόμη τώρα. Πάντω πιστεύω ότι οι περισσότεροι λογικοί παρατηρητές θα ε, θεωρήσουν ότι προσέφερε η Συμφωνία του Ελσίνκη ε, στις αλλαγέ που επισυνέβησαν στην Ανατολική Ευρώπη. Μάλιστα, σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Κύριε καθηγητά, Σάμπα, το 1975 η δήλωση του Ελσίνκη έλεγε ότι η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να συμμετάσχει σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν ένα από τα τρία περίφημα καλάθια της Συμφωνίας του Ελσίνικη. Δεν έχουμε βέβαια παρόμοια κατάσταση τώρα ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Κίνα. Δεν έχει συμφωνηθεί κάτι τι τέτοιο. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλες και όλους για την συζήτηση. για την ανταλλαγή απόψεων και τα σχόλια που ακούστηκαν στο τέλος και από τους Ευρωβουλευτάς ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Εξετάζουμε την Κίνα από διάφορες σκοπιές και μας δώσατε και πολλές απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το πώς μπορούμε να συμβάλλουμε σε αλλαγές σε μια χώρα όπως η Κίνα. Μας δώσατε πολλές συμβουλές και συστάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και απέναντι σε άλλες χώρες όπου σημειώνονται τέτοια σημαντικά προβλήματα. Νομίζω ότι καλώς χρησιμοποίησαμε το δίωρο αυτό και με την ευκαιρία θα ήθελα να καλωσορίσω τον προσκεκλημένο μας που είναι παρόν, διότι στις 3 Δεκεμβρίου είναι η Διεθνής ημέρα αναπήρων και έχουμε εδώ κοντά μας την κυρία Γέσνη Μερνίκουση η οποία εκπροσωπεί εδώ το Αιθιοπικό Κέντρο Αναπηριών και Ανάπτυξης. Η ίδια είναι ε, τυφλή, ε, έχει κάνει σπουδές νομικές και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η Σουηδική Προεδρία Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε παρούσα εδώ. Κύριε Νικούση θέλετε να λάβετε το λόγο για να πείτε λίγα λόγια. Θα ήθελα να ευχαριστώ την Πρόεδρο που μου επιτρέπει να μιλήσω για αυτή την ε, εξαιρετική σημασία εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως υπόθηκε νωρίτερα, κατάγομαι από την Αιθιοπία. Το όνομα μου είναι Νιγκούσιε. Ίσως θα σας ενδιαφέρει να ακούσετε την ιστορία μου. Τυφλώθηκα σε ηλικία 5 ετών. Στην περιοχή Εμχάρα, στην ύπεθρο της Αιθιοπίας, όπου δεν υπάρχει υποδομή και βασιζόμαστε και ασκούνται ακόμη παραδοσιακές πρακτικές που είναι πολλές φορές επικίνδυνες, όπως πρώιμος γάμος για τις κοπέλες. Η τυφλότητα, εμένα, η τύφλωση εμένα μου φάνηκε χρήσιμη τελικά, διότι κρίθηκα κατάλληλη για γάμο στην περιοχή μου, έτσι μεταφέρθηκα σε ένα αστικό κέντρο, μπόρεσα να πάω στο σχολείο, να σπουδάσω μετά στο Πανεπιστήμιο νομικά και να κάνω και μεταπτυχιακές σπουδές. Μπόρεσα λοιπόν να κερδίσω χάρη στην τύφλωση αυτήν, έστω και αν δεν είναι κάτι το οποίο θα συνιστούσε κανέναν σας. Εγώ θα μιλήσω για τις νέες προτάσεις ε, που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα. Το ε, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρίες. Όπως καλύτερα από μένα γνωρίζετε εσείς, την περασμένη εβδομάδα κυρώθηκε από την ε, Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Θα μιλήσουμε ασφαλώς και για τα Ηνωμένα Έθνη, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία είναι ένα έγγραφο, διεθνές έγγραφο για τα δικαιώματα του ανθρώπου και ως τέτοιο είναι το πρώτο του 21ου αιώνα. Τα συμβαλόμενα μέρη καλούνται να προαγάγουν και να κάνουν σεβαστά τα δικαιώματα του ανθρώπου, την ακαιρεότητα των ατόμων με αναπηρίες. Το υιοθέτησαν, το έγγραφο, το υιοθέτησε η Γενική Συνέλευση ε, του Ηνωμένων Εθνών και θα τεθεί σε ισχύ σε 12 μέρες περίπου, όταν κλείσουν δηλαδή τρία χρόνια από την έγκρισή του. Όμως είναι ένα έγγραφο το οποίο δεν προέκυψε από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάστηκαν πολλοί αγώνες, πολλές συζητήσεις, πολλές συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων που εξέταζαν και τις επιπτώσεις του. Και εμείς υπενθυμίζαμε πάντοτε το 87 η Σουηδία ήταν εκείνη η οποία είχε προαγάγει ε, και προβάλλει την ανάγκη για ένα πλαίσιο για τα άτομα, νομικό πλαίσιο, διεθνές νομικό πλαίσιο για τα άτομα με αναπηριες τωρα Ύστερα από 9-10 χρόνια δουλειά μπορέσαμε να φτάσουμε στην Σύμβαση των Εθνών που αποτελεί το πρώτο νομικά δεσμευτικό έγγραφο στα ανθρώπινα δικαιώματα σε διεθνές επίπεδο. Τι σημαίνει αυτή η σύμβαση. Ακολουθεί την παράδοση του αστικού δικαίου, έχει δηλαδή ένα προήμιο στο κόρπους, πλην όμως δεν έχει διαφορετικά τμήματα όπως ακολουθούν ε, οι άλλες, ε, όπως είναι η μέθοδος που ακολουθείται για τις άλλες συμβάσεις των ΟΕΕ. Υπάρχει το άρθρο υπαριθμών 1 το οποίο προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης, δεν ορίζει όμως τι είναι αναπηρία. Απλώς στο στόχο της σύμβασης ορίζει ε, ότι ορίζει ποια είναι τα άτομα με αναπηρίες. Ως στόχο όμως, όχι ως πεδίο. Επίση, Επίσης στα άρθρα 4 έως 32 ή μάλλον 30 αναφέρεται στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Δεν βλέπουμε να εφευρίσκονται με την σύμβαση αυτή νέα δικαιώματα για τα άτομα με αναπηρίες. Απλώς ε, εκφράζεται μία έκκληση να δοθεί περισσότερη προσοχή στα άτομα αυτά σε σχέση με τα όσα έχουν ήδη προβλεφθεί από διεθνείς συμβάσεις, έγραφα ε, για τα άτομα με αναπηρίες. Χωρίς να αρνούμαστε το γεγονός ότι εκφράζονται κάποιες περιγραφές νέων δικαιωμάτων, ε, δηλαδή το δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση και για ενσωμάτωση στην κοινότητα και το δικαίωμα στην κινητικότητα είναι δικαιώματα που για πρώτη φορά καταγράφονται, όπως επίσης και η προσβασιμότητα. Κάποιες κύριες ε, αρχές, κατευθυντήριες αρχές όπως τις αποκαλούμε, τη σύμβαση. Ε, είναι αρχές τις οποίες καλούνται να ε, ακολουθούν όλες οι χώρες. Ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια, αποφύγη των διακρίσεων, πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ενσωμάτωση στην κοινωνία, ο σεβασμό τη διαφορά, η αποδοχή των ατόμων με αναπηρίες ως ε, κομματιού της, ε, ε, της ποικιλία που παρουσιάζει το ανθρώπινο είδο, του, το δικαιώματα στη διαφορά δηλαδή, η προσβασιμότητα, η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, ο σεβασμό για την προστασία ο σεβασμός και η προστασία των, ε, της ταυτότητας και των ε, παιδιών με αναπηρίες αλλά και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Έχουμε λοιπόν, χάρη στο έγγραφο αυτό, το σεβασμό των δικαιωμάτων μας, έχουμε τη δυνατότητα να να υψώσουμε τη φωνή μας. Πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο μιλά υπέρ της ενσωμάτωσης και δεν δημιουργεί ένα νέο γκέτο των ανθρώπων με αναπηρίες. Έχουμε λοιπόν πιστεύουμε πολλά να περιμένουμε και ρόλο σημαντικό που μπορούν να διαδραματίσουν τα κράτη της διεθνούς κοινότητας. Επίσης, θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι δεν θα πρέπει όπως σε ορισμένες χώρες στην Κίνα και άλλες χώρες που έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσουν τα άτομα αυτά ως προβληματικά, ως ασθενή, ως ε, άτομα που πρέπει να μπουν στο περιθώριο. Και κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω ότι η προσφορά αυτής της Διεθνούς Σύμβασης είναι πάνω απ' όλα η συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, η δυνατότητα για ενσωμάτωση. Αυτό είναι το επίτευγμα, πάνω απ' όλα για μένα προσωπικά που είμαι άτομο με αναπηρία και η δυνατότητα που μου δίνει, η διαβεβαίωση που μου δίνει τόσο εμένα όσο και των άλλων ανθρώπων μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να μιλήσουν και δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας τους είναι αυτή η δυνατότητα ακριβώ που μας δίνει η συμμετοχή στις κοινωνίε μας. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, Κύριε Νιγκούση, για τη δήλωσή σας. Σας άκουσα με προσοχή. Σας παρακολούθησα όσο μιλούσατε και είδα να εκφράζετε μέσα από το πρόσωπό σας όχι μόνο η εμπειρία που έχετε, αλλά και η αποφασιστικότητα, η στράτευσή σας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι αγώνες σας για τα άτομα με αναπηρίες. Είναι πολύ σημαντική η δηλώση σας πιστεύω. για την προαγωγή του θέματος αυτού, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Θα κάνουμε μια συζήτηση με επίκεντρο το θέμα αυτό την Άνοιξη στην Υποεπιτροπή μας και έτσι θα έχουμε πιστεύω πιο ε, τη δυνατότητα για πιο εκτενή διάλογο, όπου θα μπορούσαμε και να αναλύσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως νομικής προσωπικότητας πλέον ε, για, την, ε, για προσχώρηση στην σύμβαση. Και τώρα περνάω στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης που έχει τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή. Ερωτήσεις που έχουν διατυπώσει οι ευρωβουλευτές και ξεκινούμε με την κατάσταση των χριστιανών στην Λιβύη. Στην Ινδία, συγγνώμη. Η πρώτη ερώτηση αναφέρεται στην κατάσταση των χριστιανών στην Ινδία. Η δεύτερη την ε, ε, περιβαλλοντική καταστροφή του Μποπάλ του 1984. Για την πρώτη ερώτηση, κατάσταση των χριστιανών και τι προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιώσει ή να ελαφρύνει τις ε, δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν, θα ήθελα να πω από την αρχή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε υπόψη των Ινδών εταίρων την ανησυχία που ε, υφίσταται στην Ευρώπη και τη βλέπουμε και από πολλές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις σχετικά με την βία και τους διωγμούς σε βάρος πολλών ευάλωτων ομάδων, περιλαμβανομένων των χριστιανών. Και είπαμε πόσο αναγκαίο είναι, εξηγήσαμε πόσο αναγκαίο είναι να προστατευτούν όλες οι ευάλωτες ομάδες, περιλαμβανομένων των χριστιανών και άλλες ομάδες όμως, όπως γυναίκες, μειονότητες, παιδιά. Εκφράσαμε την ανησυχία μας αυτή και επισήμως θέσαμε δηλαδή ε, το θέμα υπόψη των ινητικών αρχών κατ' επανάληψη στον διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδιών που γίνεται κάθε χρόνο στο Δελχή. Το θέσαμε και υπόψη της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ινδία και το 2008 στην διάσκεψη κορυφή στη Μασαλία μεταξύ Ένωσης και Ινδιών και στις προπαρασκευαστικές συναντήσεις αλλά και στο υψηλότατο επίπεδο όπου και ο ίδιος ο Πρωθυπουργό ΣΥΝΚ δέχθηκε ε, ότι υφίσταται ε, το πρόβλημα αυτό και ότι λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση του. Η κατάσταση κυρίως αναφέρεται στους χριστιανούς της Νουρίσα που ε, είδε το φως της δημοσιότητας και πριν από λίγα χρόνια και που ασφαλώς ανησυχεί και τους επικεφαλής της εκπροσώπησης της Ένωσης στην ε, στις Ινδίες και που προδιετίας οργάνωσαν μια εξεταστική ε, αποστολή ε, στην, περιοχή αυτή. Η ίδια ομάδα, δηλαδή οι Heads of Mission, οργανώνουν και συναντήσεις με μη κρατικές οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Νουρίσα για να εξετάσουν τι άλλο μπορεί να γίνει, ποιες πιέσεις μπορούν να ασκηθούν προς την κατεύθυνση μιας βελτίωσης της κατάστασης. Τελευταίο σχόλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για προτάσεις με προτάσεις που θα υποβληθούν μέχρι με προσφορές που θα υποβληθούν μέχρι τέλους Ιανουαρίου για την παροχή υπηρεσιών ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη όλων και ευαλώτων ε, ε, ομάδων όπως γυναίκες, μειονότητες και ε, θρησκευτικέ μειονότητε, γιατί αυτό είναι και μια εκδήλωση του ενδιαφέροντος που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα και η ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανθρώπινα δικαιώματα στο Δελχή επίσης εξετάζει ειδικά το θέμα αυτό της κατάστασης των μειονοτήτων. Και αν με επιτρέπετε να προχωρήσω αμέσω στην δεύτερη ερώτηση. Ο Προεδρεύων. Θα ήθελα ο συντάκτης της ε, ερώτησης, εάν έχει κάποιες ε, συμπληρωματικές ερωτήσεις, να τη θέσει ο κ. Στόκος. Νομίζω όμως ότι δεν έχει τίποτε να προσθέσει στην ερώτηση. Είμαι παρόν ε, κύριε Πρόεδρε, παρόν λέει ο κ. Στόκος. Σας ευχαριστώ για την απάντηση που δώσατε Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόβλημα είναι το ίδιο κατά τη γνώμη μου και στην περίπτωση αυτή όπως και στην περίπτωση της Κίνας. Δηλαδή, εννοώ ότι η σιωπηλή ε, διπλωματία θα ήθελα να γνωρίζω πόσο βοηθεί στην περίπτωση αυτή, πόσο συμβάλλει. Τι χρειάζεται να γίνει για να τεθούν τα θέματα αυτά εντονότερα. Καθώς προέρχομαι από πρώην κομμουνιστική χώρα, γνωρίζω από προσωπική εμπειρία ότι τα θέματα δεν ετίθετο πάντοτε επί εποχής Τσαοσέσκου. Δηλαδή, ναι, μεν έθεταν κάποιες ερωτήσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι ευρωπαϊκές χώρες και μετά Όλοι, όλοι ησύχαζαν ε, διότι θεωρούσαν ότι είχαν τεθεί τα θέματα και τα πράγματα συνέχιζαν να εξελίσσονται με τον ίδιο τρόπο και τότε στη Ρουμανία όπως τώρα άλλωστε στην ε, Κίνα ή στις Ινδίες. Δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ανελευθερία άσκησης ε, ε, της θρησκείας και ούτω καθεξής συνέχιζαν με τον ίδιο τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ή οι Ηνωμένε Πολιτείες έχουν αν είχαν, αν είχαν δραστηριοποιηθεί εντονότερα τότε στην περίπτωση της Ρουμανίας, νομίζω ότι ο Τσαουσέσκο εν τέλει θα είχε υποχωρήσει. Γι' αυτό ρωτώ αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κάνει κάτι το πιο αποτελεσματικό. Για παράδειγμα, για το νόμο, για το γλωσσικό νόμο στην Σλοβακία. Η προσέγγιση στερείται βάσης γνώσης από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Να πρόκειται στην πραγματικότητα για μια έντονη κατάφορη παραβίαση των γλωσσικών δικαιωμάτων στην περίπτωση της Σλοβακίας. Τι είδους αξίες υποτίθεται ότι εκπροσωπούμε όταν δεν υπερασπιζόμαστε παρκώς τέτοιες διοκόμενες ομάδες όπως ε, μουσουλμάνους ή και χριστιανούς. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Προεδρεύων και Τόκες και ας έρθουμε τώρα στην ερώτηση της Μπάρμπαρα Λόχ Μπίλερ σχετικά με την κατάσταση στο Μποπάλ μετά από εκείνη την ε, γνωστή περιβαλλοντική καταστροφή του 1984. Θα ήθελα καταρχάς να πω η Επιτροπή ανησυχεί ακόμη ιδιαίτερα για την ε, ανθρωπιστική και ιατρική διάσταση του ατυχήματος του Μποπάλ. Δεν έχουμε όμως, όπως δεν είχαμε και το 84, μέσα στη διάθεσή μας επαρκή ώστε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση ή να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Βέβαια θα μπορούσε κανείς να προβάλλει το επιχείρημα ότι θα έπρεπε να έχουμε ε, προσφέρει τεχνική αρρωγή για, την, ε, για το καθαρισμό της περιοχής, για την εξασφάλιση πόσιμου καθαρού, πόσιμου νερού, για τον πληθυσμό της περιοχής. Και σε αυτό ε, θα απαντήσω ότι μόνο σε αίτημα της Συνδικής Κυβέρνησης θα μπορούσαμε να έχουμε ανταποκριθεί. Το 2004 με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχαμε ήδη ένα πρόγραμμα συνεργασίας με σημαντική χρηματοδότηση, το οποίο όμως εξορισμού πρέπει να είναι προσδιορισμένο με στόχους συγκεκριμένους και εγκεκριμένους από τις κυβερνήσεις, από την κυβέρνηση, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, όπως είχε γίνει. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό εστιαζόταν ουσιαστικά στους κοινωνικούς τομείς, την υγεία, την εκπαίδευση και δεν κάλυπτε ε, άλλες δραστηριότητες, ούτε επέτρεπε την επέκτασή τους σε δραστηριότητες διαφορετικές, όπως στην περίπτωση του Μποπάλ. Και μάλιστα δεν υπέβαλε σχετικό αίτημα και η κυβέρνηση της Ινδίας. Τούτων λεχθέντων, και έχοντας υπόψη την ανάγκη να προσφέρουμε αρρωγή στην Ινδία σε περίπτωση τέτοιων μεγάλων καταστροφών και ατυχημάτων, Έχουμε διαπραγματευτεί και προσφέρει στην ειδική κυβέρνηση 10 εκατομμύρια ευρώ για το 2004 για ένα εσωτερικό πρόγραμμα της ειδική κυβέρνηση, δηλαδή πρόγραμμα διαχείρισης καταστροφών και ατυχημάτων, το οποίο αναπτύσσει συνεργασία με το ε, πρόγραμμα ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, η ειδική κυβέρνηση. Σε κάθε επίπεδο, εθνικές, από την εθνική κυβέρνηση, τις περιφερειακές, αλλά ακόμη και την τοπική αυτοδιοίκηση, ακόμη και στο επίπεδο του χωριού αναπτύσσεται το πρόγραμμα αυτό και μπορεί να εστιάζεται κατά κύριο λόγο στις φυσικές καταστροφές, ωστόσο επειδή έχει περιγραφεί ως ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει να αντιμετωπίσει τις ε, ανάγκες μιας συγκεκριμένη κοινότητας ε, σε μια περίπτωση καταστροφής, σαφώς υποδεικνύει, πιστεύω, την ανάγκη την οποία αισθάνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφέρει την υποστήριξή της και σε τέτοιου είδου προβλήματα που οφείλονται σε συγκεκριμένε δραστηριότητες. Επίσης, δε, σημειώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει, όπως εδώ και χρόνια συμμετέχει, σε ένα περιβαλλοντικό διάλογο με τις ινδικές αρχές σε πολλά επίπεδα, διάφορα επίπεδα που φτάνουν μέχρι το Υπουργικό, όπου έχουμε και ανταλλαγή απόψεων και διάλογο τακτικό και εξέταση ενός ευρύτατου φάσματος περιβαλλοντικών θεμάτων όπου πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να προσφέρει προσθέμενη αξία στην Ινδία και εδώ έχουμε να κάνουμε και με την περιβαλλοντική νομοθεσία και με πολλά άλλα διάφορα θέματα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτός ο διάλογος και αυτές οι ανταλλαγές απόψεων και στις μεταρρυθμίσεις συμβάλλουν και βοηθούν τους Ινδούς να εισαγάγουν, ε, να αντιληφθούν καταρχάς ότι υπάρχουν διαφορετικά ρυθμιστικά συστήματα, κανονιστικά συστήματα και να εισαγάγουν εν τέλει εκείνα τα οποία θεωρούν ε, πιο χρήσιμα. από την εποχή αυτή τη καταστροφή του Μποπάλ, επίση έχει η Κίνα εισαγάγει πολύ αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία που στόχο έχει να αποτρέψει επανάληψη τέτοιων ατυχημάτων. Θα ήθελα επίση να αναφέρω ακόμη δύο λόγια για το ζήτημα τη εταιρική ευθύνη. Τη ευθύνη δηλαδή ευρωπαϊκών εταιριών ή εμπορικών επιχειρήσεων οι οποίε δραστηριοποιούνται στην Ινδία. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο ε, γύρθη στον διάλογο με τους ε, Ινδούς στα θέματα απασχόλησης και εμπορικών σχέσεων από την αντίστοιχη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, μάλλον θα, γίνει κάποια, θα υπάρξει κάποια εξέλιξη ως προς το ζήτημα της εταιρική ευθύνη και της ευθύνη των εμπορικών επιχειρήσεων, πολύ πιο ουσιαστική δηλαδή για το μέλλον. Δεν πρέπει όμως και να λησμονούμε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο διαπραγματεύσεων μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Ινδία. και έχουμε δεσμευθεί στη διαπραγμάτευση ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου με τους Ινδούς ε, για την ε, ανάπτυξη, την εμπορική ανάπτυξη που θα κάλυπτε και τις εμπορικές πτυχές αλλά και τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οποιαδήποτε άλλη πτυχή μιας τέτοιας εμπορικής συμφωνίας ή συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών. Αυτό πάντα σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και πιστεύω ότι είναι μια διάσταση η οποία εγγράφεται πιστά μέσα στις ε, προτάσεις και για την παγκοσμιοποίηση με την αίτηση ανταγωνιστικότητας αλλά και της βιωσιμότητας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πώς θα ήθελε της ερώτησης να απαντήσει, κυρία Σας ευχαριστώ για την πολύ απάντηση. έχω όμως μία ερώτηση. Ε, εάν στη με την ε, Ινδική κυβέρνηση, μέσα στο διάλογο που αναπτύσσεται, έχετε ζητήσει από την Ινδική κυβέρνηση να συστήσει μια επιτροπή ερευνητική του ατυχήματος της Μποπάλ με τους κατάλληλους φόρους και το προσωπικό, πράγμα το οποίο ζητούν διακάως οι κάτοικοι της περιοχής. Επίσης, πέρυσι ο ειδικός συζητητής των ΗΕ Εθνών για τις σχέσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με, το την προστασία των δικαιωμάτων υπεγράμισε ιδιαίτερα για την Ινδία ότι χρειάζεται να προστατευτούν, να αναγνωριστούν και να προστατευτούν τα δικαιώματα των θυμάτων, των παραβιάσεων ανθρωπινών δικαιωμάτων και ότι η ενίσχυση της δέσμης των δικαιωμάτων και μέσα από τις εμπορικές σχέσεις, τις σχέσεις συναλλαγών με μεγάλες εταιρείες όπως χημικής ε, βιομηχανίας, ε, ιδιαίτερα έχουν συμβάλει στην ε, προαγωγή των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Λόχμπίλερ στο επόμενο ερώτημα η κυρία, της κυρίας Ελίζαμπετ Γέκλε, κατάσταση στο Βιετνάμ. Μοναχοί και μοναχές, παρακαλώ. O, widzę tutaj jest przedstawiciel komisji, który w tej sprawie zechce odpowiedzieć. Proszę bardzo. Thank you, Mr. Chair. Uh, well, I would like to stress that the Commission and Member States... Εγώ τονίζω ότι και η Κομισιόν και οι χωρισμένοι γνωρίζουν την κατάσταση στην Μονή Μπάτνια. Ε, δεχθήκαμε διάβημα 10 μοναχών από την Μονή για να, αλλάξουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις μεταξύ τους για την κατάσταση στην Μονή. Στις 11 Νοεμβρίου η επικεφαλής των αντιπροσωπιών της Ένωσης Πρέσβης δηλαδή στο Ανόη συναντήθηκαν με τον αρμόδιο υπουργό στο Ανόη για να εκφράσουν τις ανησυχίες ε, της Ένωσης για τις απειλές ε, που, έχουν, που έχει υποστεί η μοναστική κοινότητα και ζήτησαν να, από τις βιετναμικές αρχές να μην φύγουν οι μοναχοί και να τους επιτραπεί να συνεχίσουν τις ειρηνικές του δραστηριότητες. Οι εκεί τώρα σκέπτονται να κάνουν μια επιτόπου επίσκεψη στην Μονή για να αξιολογήσουν την κατάσταση. Στην βάση δε της αναφοράς που θα υποβάλουν θα αποφασιστεί η περαιτέρω δράση. Το θέμα είναι στην ατζέντα της επόμενης, ε, του επόμενου γύρου του διαλόγου ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ που θα γίνει ε, μέσα Δεκεμβρίου στο Ανόη και γνωρίζουμε και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε την επόμενη εβδομάδα για τα θέματα αυτά και που ρίχνει ακόμη περισσότερο φως στην υπόθεση αυτή. Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση του Βιετνάμ θα επανεξετάσει την θέση της στο θέμα αυτό. Mm, Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γέγλε. Θέλετε να σχολιάσετε. Δεν τα σχολιάσετε περισσότερο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ και, τις, και τους συναδέλφους μου για την υποστήριξη που έδωσαν στο ψήφισμα την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Συζητήσαμε σήμερα πολλά θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι μέγα το καθήκον αυτό. Ευχαριστώ για όλα όσα θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε μαζί και για το θέμα αυτό αλλά και για πολλά άλλα. Ας προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα, στην επόμενη ερώτηση που θέτει η κυρία Νικόλ Νίλσεν για την πρόσβαση στο νερό στα πλαίσια της ισραλο παλαιστινιακης σύγκρουσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε. Πρόσβαση προϊόντων από τα Παλαιστινιακά εδάφη. Η βασική αρχή που ισχύει στον τομέα αυτό, αν και βέβαια κυρίως ε, ενδιαφέρεστε για, το νέο, για τη νέα συμφωνία για τα αγροτικά προϊόντα. Οι γενικές αρχές λοιπόν είναι ότι η κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, θεωρεί την Συμφωνία Συνδέσεως μεταξύ Ενώσεως και Ισραήλ αφορά αποκλειστικά διακόπτη κάποιος. Δεν, ακούω, δεν ακούγονται φαίνεται όλες οι μεταφράσεις. Παρακαλείτε σε μια στιγμή να περιμένετε να δουν όλοι οι διερμηνείς ότι έχουν όντως πατήσει τα κομβία. Λοιπόν, για να ανοίξω τα μικροφωνά του. Έλεγα λοιπόν, συνεχίζει ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπενθύμιζα μάλλον τι βασικέ αρχέ ό,τι αφορά την πρόσβαση προϊόντων από τα κατεχόμενα εδάφη. Οι αρχέ αυτέ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η συμφωνια Συνδέσεω Συνδέσεως Ένωση εφαρμόζεται αποκλειστικά στο έδαφο τη επικράτεια του κράτου του Ισραήλ, όπω αναγνωρίζεται από την διεθνή κοινότητα σύμφωνα με τα οικία ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ενωμένων Εθνών. Δηλαδή, προϊόντα τα οποία προέρχονται από Ισραηλινούς επικισμούς δεν ε, μπαίνουν στις προτιμησιακές, στην προτιμησιακή μεταχείριση όταν έρχονται στο, στην επικράτεια της κοινότητας. Αυτό περιλήφθηκε και στην νότης του Importers που ε, ήδη ε, δημοσιεύθηκε το 2005 ε, στο επίσημο έντυπο της κοινότητας. Και κυρίως για τη νέα συμφωνία για τα αγροτικά προϊόντα και την περαιτέρω απελευθέρωση αγροτικών αλλιευτικών προϊόντων, συμφωνία η οποία υπογράφηκε στις αρχές Νοεμβρίου και πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2019. νέα αυτή συμφωνία βασίζεται στις αρχές που μόλις ανέπτυξα προηγουμένως. Και ως εκ τούτου τα προϊόντα αυτά, δηλαδή αγροτικά και αντιευτικά προϊόντα, καλύπτονται από τη συμφωνία αυτή και εφόσον προέρχονται από ε, Ισραηλινούς επικισμούς, δεν εισέρχονται στο καθεστώς ε, προτιμησιακής μεταχείρισης. Η άλλη ερώτηση αναφέρεται στο νερό. Και ιδιαίτερα αναφέρεται σε μια έκθεση που εξέδωσε η Διεθνής Αμνηστία για το θέμα του νερού στα κατεχόμενα εδάφη. Η Κομισιόν γνωρίζει βεβαίως την έκθεση, είχαμε και επαφές με τη Διεθνή Αμνηστία, γνωρίζουμε το περιεχόμενο της εκθέσεως και το εξετάζουμε, διότι μόλις το δημοσιεύθηκε η Ρίστον Παρόδο. Το ε, εξετάζουμε λοιπόν προσεκτικά το περιεχόμενο της ε, έκθεσης αυτής. Σε ό,τι αφορά τώρα το ρόλο του νερού και ε, των αποχαιρετικών συστημάτων κτλ. μέσα στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Η χρήση του νερού και, και για ε, χρήση του νερού δηλαδή καθαρά αλλά και οι αποχαιρετεύσεις είναι ε, δικαίωμα το οποίο εντάσσεται μεταξύ των υπολείπων δικαιωμάτων μέσα στον κώδικα, στο Διεθνή Κώδικα ε, Πολιτιστικών και Άλλων Δικαιωμάτων, στο άρθρο 11. Και όλα αυτά εξασφαλίζουν ένα επαρκές ιδιωτικό επίπεδο. Αυτό το νόημα έχει. Υπάρχει και ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών για το νερό και τις ε, αποχετεύσεις, τα οποία έχουν ε, ψηφιστεί και από το Σύμβολο Ασφαλείας. Συμμετέχει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ακολουθούμε τις συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων. Σε ό,τι αφορά τώρα συγκεκριμένα το δικαίωμα χρήση του νερού στην περιοχή αυτή, η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι υπάρχουν προκλήσει σε ό,τι αφορά την ε, χρήση, πρόσβαση και διαχείριση των υδάτινων πόρων ε, μεταξύ Ισραήλ και κατεχόμενων εδαφών. Αυτέ οι προκλήσει έχουν βέβαια και επιπτώσει και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Για παράδειγμα, για θέματα μη διακρίσεων και για συμμετοχή στην διαχείριση του νερού. Η πολιτική μας είναι διαρκής. Ενθαρρύνουμε το Ισραήλ και τους γειτονέ του να θέσουν τα θέματα του νερού και να συμπεριληφθούν αυτά στις συνολικές διαπραγματεύσεις. Άλλο θέμα το οποίο έθιξε η αξιότιμη βουλευτής και πιο συγκεκριμένα τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποστηρίξει προγράμματα ανάπτυξης στον τομέα αυτό υπάρχουν, υπάρχει ένας αριθμός προγραμμάτων τα οποία υποστηρίζονται χρηματοδοτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα η Περιφερειακή Τράπεζα Δεδομένων για το νερό που περιλαμβάνει τις αρχές του Ισραήλ, της ε, Παλαιστινιακής Αρχής, της Ιορδανίας για την χρήση δηλαδή των δεδομένων σχετικά με το νερό. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια και ιδίως να συμβάλλουμε στην ελάφρυνση των προβλημάτων και δυσχεριών και κυρίως για την λωρίδα της Γάζας. Θα συνεχίσουμε, διότι αυτή ήταν πάντοτε η πολιτική μας, να πιέζουμε το Ισραήλ να ελαφρύνει τους ε, μεθοριακούς περιορισμούς και να επιτρέψει την δίωδο υλικών και εξοπλισμού για την βελτίωση της παροχής νερού. Η Κομισιόν επίσης θα συνεχίσει να προσφέρει χρηματοδότηση για έργα βελτίωσης της παροχής νερού και των αποχετεύσεων. Η πολιτική μας είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί με την Παλαιστινιακή Αρχή για να προσφέρουμε χρηματοδότηση και για την Δυτική Όχθη για, για συστήματα παροχής νερού, άρδευσης γεωργικών γεών και αποχέτευσης. Θα εξετάσουμε το θέμα να θέσουμε το πρόβλημα αυτό και στον πολιτικό διάλογο με το Ισραήλ, όπως κάνουμε άλλωστε μέσα στα πλαίσια της πολιτικής γειτονίας. E, ευχαριστώ πολύ. η να Ευχαριστώ για αυτές τις απαντήσεις. Αλλά εγώ δεν ε, αισθάνομαι σίγουρη για το θέμα της ε, ανιχνευσιμότητας των προϊόντων που εισάγονται από το Ισραήλ. Ξέρουμε ότι στα καφάσια των φρούτων όλα είναι ανακατεμένα. Ε, αντιαπικιοκρατικές Ισραηλινές οργανώσεις κάνουν έρευνες ε, σχετικά με αυτό. Έχουν και βάσεις δεδομένων επίσης σχετικά και εργάστηκαν γύρω από χίλιες επιχειρήσεις οι οποίες κερδοσκοπούν με την απεικιοκρατία. Και πολλά στοιχεία τα έχουμε και στις ιστοσελίδες αυτών των οργανώσεων. Οι επιχειρήσεις Εόλια, Δέξια και Αγκρέσκο, η οποία είναι κρατική επιχείρηση, στον Ιορδάνη, στην περιοχή του Ιορδάνη, έχει το 60% των εξαγωγών στα χέρια της και το μεγαλύτερο ποσοστό είναι Παλαιστίνοι εργάτες που εργάζονται με χείριστες συνθήκες και χαμηλότατους μισθούς, χαμηλότερους από αυτούς που παίρνουν οι Ισραηλινοί Και πολλά από τα προϊόντα έχουν ετικέτες προϊόντα Παλαιστίνης. Και αυτό για να γίνει εισαγωγή σε χώρες οι οποίες απαγορεύουν την εισαγωγή Ισραηλινών προϊόντων. Διότι σήμερα το κίνημα ταρίσματος των Ισραηλινών προϊόντων είναι σημαντικό. Οι Παλαιστίνοι έχουν ξεκινήσει αυτό το μποϊκότ, έχουν απευθύνει έκκληση και ζητούν να ασκείται μποϊκότ προς αυτά τα προϊόντα τα οποία παράγονται με κάκιστες συνθήκες χωρίς το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απαιτείται λοιπόν μια πραγματική πολιτική βούληση και να κοιτάμε από πού προέρχονται οι χορμάδες, τα σίκα, οι ντομάτες κλπ. Ευχαριστώ. Η απάντηση της Επιτροπής φαίνεται πως δεν ικανοποίησε την κυρία Κιλ Πρέπει λοιπόν να συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα αυτό η Επιτροπή.